Good Καλό σας απόγευμα αγαπητές και αγαπητοί φίλοι. Αν δεν έχετε ενστάσεις για την ημερησία διάταξη τότε θεωρείτε εγκεκριμένη και θα ήθελα να κάνω ορισμένε ανακοινώσει και πρώτα το γλωσσικό μας καθεστώς. Μας λείπουν σήμερα τα γοεδελικά και τα κροατικά. Οι, ε, στάσεις, το, ε, συγγνώμη, οι των συντονιστών ε, θα πρέπει να εγκριθούν. Έχουμε πρώτα Γκυγιόμ S&D Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για το βαθμολόγιο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την δικαιοσύνη, αν ε, δέχεστε την πρόταση αυτή. Κύριε Ζιρέ, έχετε διαδικαστικό. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Για τις 5 η ώρα είναι προγραμματισμένη ψηφοφορία για νέο σχέδιο ψηφίσματο για την Πολωνία. Όμως δεν προβλέπεται στο σχέδιο ημερησία διατάξεω συζήτηση και πέραν αυτού είναι ασαφές και ποιε είναι οι προθέσεις πίσω από αυτό το σχέδιο. Εγώ διάβασα το σχέδιο και αυτό παραπέμπει σε συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την κίνηση του άρθρου 5 κατά της 7, ε, κατά της Πολωνίας, που προβλέπει όμως ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο όταν ε, θα υπάρξει η ενισχυμένη πλειοψηφία. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί άραγε σήμερα έρχεται σε ψήφιση η, το σχέδιο αυτό ψηφίσματος, ενώ δεν προβλέπεται συζήτηση. Η πρότασή μου λοιπόν, λοιπόν είναι να αφαιρεθεί από την ημερησία διάταξη, να διευκρινιστεί πρώτα η κατάσταση, εάν δηλαδή υπάρχει πραγματικά λόγος. Και να δούμε αν όντως θα πρέπει να τεθεί ε, επιτάπητο στο θέμα αυτό στο μέλλον κάποια στιγμή. Αυτό το έχω στο υπαριθμό 4 των ανακοινώσεων μου, την ηλεκτρονική ψηφοφορία δηλαδή αργότερα σήμερα, που γίνεται μετά από αίτηση των συντονιστών, την απόφαση των συντονιστών αυτή, ώστε να έχουμε την έγκριση για να πάμε στην Ολομέλεια. Δηλαδή πρόκειται για ψηφοφορία τεχνικού χαρακτήρα που θα μας επιτρέψει να μεταβούμε με το σχέδιο αυτό στην Ολομέλεια, διαδικασία την οποία οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Για το λόγο αυτό δεν προβλέπεται συζήτηση και γι' αυτό θα παραμείνει στην ημερησία διάταξη και θα κάνουμε αυτή την μοναδική ψηφοφορία, ενιαία ψηφοφορία χωρίς συζήτηση. Και πρόκειται για ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άλλωστε έχετε ενημερωθεί εγκαίρως όπως και όλες οι πολιτικές ομάδες και ο συντονιστής σας. Και η πλήρη συζήτηση βεβαίως θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ όμως που θέσατε το θέμα. Όπως έλεγα, η ηλεκτρονική ψηφοφορία στην οποία αναφέρεται ο κύριος Γιούρεκ θα διεξαχθεί στις 5 η ώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 5 το απόγευμα και στις 19 και 45 προβλέπεται κοινή συνεδρίαση Λίμπε Έκον. Και στις 6.30 θα τη συζήτηση για την νομοθεσία, για πρόταση νομοθεσίας για το 1665 μάλλον 2000, για τον κανονισμό 2016 κάθετος 1675. Άρα τώρα έχουμε το θέμα 3 της σημερινής διάταξης και ευχαρίστως υποδέχομαι τον Επίτροπο κύριο Κίνγκ εισαγωγικά για το θέμα αυτό υπενθυμίζω ότι οι επίτροποι Κίνγκ και Αβραμόπουλος στις 2 έκτου ανακοίνωσαν την ίδρυση Επιτροπής για την ριζοσπαστικοποίηση στα πλαίσια μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσίασε στις 7 Σεπτεμβρίου ο κ. Κίνγκ σύμφωνα με μια γαλλογερμανική ιδέα για τη δημιουργία ενός κέντρου για τη μελέτη της ριζοσπαστικοποίησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε γίνει στο Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2017, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ε, συστήσει την Επιτροπή αυτή με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τις χώρες μέλη, από άλλους οργανισμούς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Επιτροπή Εξωτερικής Δράσεως και ε, με εκπροσώπους του συντονιστού κατά της τρομοκρατίας και η δική μας επιτροπή συμμετέχει ως παρατηρητής. Υπάρχει προσωρινή έκθεση τώρα που περιλαμβάνει τα πρώτα ευρήματα κάθε του πορίσματα σήμερα και πολύ ευχαρίστως θα ακούσουμε τον ε, Επίτροπο κύριο Κίνγκ που θα αναπτύξει τα ε, πρώτα αυτά ε, πορίσματα της Επιτροπής. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου συνίσταται στο ότι έχει συζητήσει ήδη στην Ολομέλεια. Χρειάζονται να γίνουν περισσότερα πράγματα για να αυξηθεί ο συντονισμό με συμμετοχή των ενδιαφερμένων μερών στον τομέα αυτό. Πολύ ευχαρίστω να δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Επίτροπο για να μπορέσει να προβεί στην παρουσίαση του θέματος. Ευχαριστώ για την έλευσή σας κύριε Επίτροπε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου προσφέρετε να προβώ σε ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα της συγκράτησης της ριζοσπαστικοποίησης και ιδίως για την ομάδα εμπειρογνωμόνων που ακούσατε μόλις τα της ιδρύσεώς της από τον πρόεδρο σας. Νομίζω ότι μαζί έχουμε ε, σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας τους τελευταίους μήνες και χρόνια. Έχουμε κάνει βήματα για την βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά και για την μείωση του χώρου όπου μπορούν να αναπτύξουν δραστηριότητα οι τρομοκράτες. Ένα απολύτως κέριο σημείο της ε, αντιμετώπισης της πρόκλησης είναι ε, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του. Δηλαδή να τηθεί το ερώτημα τι κάνει κάποιον ο οποίος έχει γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ, στην Ευρώπη, να καταλήξει στην χρήση βιώτατων ε, μεθόδων. Έχουν, υπάρχουν πολλές, ε, πολλές πρωτοβουλίες σχετικά. Υπάρχει το δίκτυο για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ριζοσπαστικοποίηση με συμμετοχή από κοινωνικού λειτουργού έω οχρονιστικού υπαλλήλου έω δασκάλου κλπ. Αυτό που χρειάζεται είναι να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στι επιτυχεί αυτέ προσπάθειε ω θεμέλια. Χρειάζεται ακόμη να περιλάβουμε και άλλου στην προσπάθεια αυτή ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις, σημαντικέ, καθώς και ερευνητές. Ορισμένοι προτείνουν, όπως υπενθύμησε ο πρόεδρός σας, τη δημιουργία νέων δομών για τον συντονισμό του έργου αυτού, όπως το κέντρο αντιρίζοσπαστικοποίησης. Στην βάση αυτού του ιστορικού, λοιπόν, συντέθηκε και η Επιτροπή και εξέδωσε την προσωρινή της έκθεση τον Σεπτέμβριο με σημαντική υποστήριξη του Συμβουλίου η έκθεση περιλαμβάνει φιλόδοξε συστάσεις και δείχνει ένα προσανατολισμό, δείχνει μια πορεία προς τα, εξής, εμπρός. Με την υποστήριξη της έκθεσης την οποία εγκρίναμε την προηγούμενη εβδομάδα, έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών για τα πιο βασικά στοιχεία των συστάσεων της προσωρινής αυτής έκθεσης και κάποιες από τις πρώτες μας απαντήσεις στις παρατηρήσεις της εκθέση αυτής, καθώς επίσης βέβαια και να ακούσω και να σημειώσω τις δικές σας απόψεις για το πώς θα προχωρήσουμε. Το βασικό θέμα το οποίο διέρχεται ως ερυθρό νήμα μέσα από όλη την προσπάθεια αυτή είναι η ανάγκη να αναπτυχθούν περισσότερες ικανότητες στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποστήριξη και παροχή βοήθεια στις χώρες μέλη για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης με ισχυρότερες μεθοδολογίες αναλύσεως, έρευνα, εκπαίδευση, ε, παροχή ε, κατευθύνσεων και βεβαίω και πρόσκληση και προς τους έξω να βοηθήσουν. Η ανάγκη αύξηση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλειών και μεταξύ των ενδιαφερμένων μερών που εργάζονται στον τομέα αυτό, να βελτιώσουν την έρευνα και την ανάλυση και να αναπτύξουν περαιτέρω πολιτικές που να βασίζονται σε συγκεκριμένες ενδείξεις οι συστάσεις της ε, ομάδας εμπειρογνωμόνων τονίζει ορισμένες από τις ε, πιο θεμελιώδεις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Πρώτα για τις φυλακές, όπου οι φυλακές μπορούν να αποτελέσουν και το εκολαπτήριο, ας πούμε, για την ριζοσπαστικοποίηση, διότι στο κλειστό περιβάλλον των φυλακών οι ορισμένοι από αυτούς ε, που ε, είναι επιρρεπείς σε τέτοια θέματα μπορεί να ε, καταστούν, να ριζοσπαστικοποιηθούν. Έχουμε και τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές, αλλά και για θέματα αποκατάστασης και επανένταξης στις κοινωνικές δομές μέσα σε όλες τις χώρες μέλη. Χρειάζεται βέβαια να ανταλλάξουμε και τις βέλτιστες πρακτικές για την εκπαίδευση του σοφρονιστικού προσωπικού και πώς ε, να αντιμετωπιστεί επιστημονικότερα η ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές. Εμείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθούμε τις συστάσεις αυτές, τις θέτουμε υπόψη των κυβερνητικών ε, εθνικών αρχών, βεβαίω συνεργαζόμαστε και με τη Βουλγαρική Προεδρία, αλλά συνεργαζόμαστε και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, του stakeholders δηλαδή, και στις φυλακές, στα σοφρονιστήρια και ε, τους άλλους συναρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Ε, για τα τέλη Φεβρουαρίου οργανώνουμε διάσκεψη με συμμετοχή δικαστών, εισαγγελέων, σοφρονιστικού προσωπικού και ε, αξιωματούχων που παρακολουθούν τα πρόσωπα που απολύονται από τις φυλακές υπό όρους και ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθεί πρόοδος και προβλέπονται και θέματα χρηματοδότησης. Θα δώσουμε και περισσότερες επιχορηγήσεις μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Justice για την ε, εκπαίδευση δικαστών. Το δε δίκτυο κατά της ριζοσπαστικοποίησης διεξάγει εκδηλώσεις με συμμετοχή προσώπων που ασχολούνται στην πράξη με το θέμα αυτό, με στόχο την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών σε συνεργασία με οργανισμούς όπως ο ΟΑΣΕ και το ε, Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, Δικαστικών Οργανώσεων. Αυτές όλες οι προσπάθειες θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τους βίους ριζοσπαστικοποιηθέντες ε, δράστες και άλλα ζητήματα ριζοσπαστικοποίησης, να καλύψουμε ευρεία ζώνη θεμάτων, μεταξύ άλλων ε, ανάλυση του κινδύνου, αλλά και τον ρόλο των θρησκευτικών ηγετών στην ριζοσπαστικοποίηση. Διερευνούμε και την ιδέα να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα ε, αξιολόγησης ισοτήμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο εμπειρογνώμονες από χώρες μέλη να αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο μεμονωμένες χώρες μέλη οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο δίκτυο αυτό, αντιμετωπίζουν θέσματα ριζοσπαστικοποίηση της φυλακές. Η έκθεση σημειώνει επίσης την πρόκληση της ανάγκης να παρασχεθεί βοήθεια και σε παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε ριζοσπαστικοποιημένα περιβάλλοντα. Το ζήτημα των επανερχομένων μαχητών, για παράδειγμα, ασφαλώς και έχει προκαλέσει συζήτηση σε όλες τις χώρες μέλη, το πώς τους παρακολουθεί η ποινική δικαιοσύνη, η ειδική προστασία που χρειάζονται γυναίκες και παιδιά. Έχουμε και εδώ ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τον αριθμό των άνω 5.000 ε, μαχητών που έφυγαν από την Ευρώπη και που από αυτούς επανέρχονται, υπάρχει όμως και ένα σημαντικός αριθμός παιδιών, τα οποία είτε μετέβησαν και αυτά εκεί, στο Ιράκ και τη Συρία, ή γεννήθηκαν εκεί και τα οποία έχουν υποστεί Πραγματικού ε, ψυχολογικού τραυματισμού, έχοντα παρακολουθήσει εκτελέσει, βασανιστήρια ή καμιά φορά μάλιστα σε πιο ακραίε περιπτώσει, εξαναγκάστηκαν ε, να προβούν σε βίαιε πράξεις τα ίδια. Και τα επιστρέφοντα παιδιά αποτελούν μια συγκεκριμένη πρόκληση την οποία δεν πρέπει να υποτιμήσουμε. Όπω συνιστά η ομάδα εμπειρογνωμόνων πρέπει να γίνει μια περαιτέρω ανάλυση σχετικά με τις προσεγγίσει όλων των χωρών μελών σε ό,τι αφορά την ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων και πιο συγκεκριμένα τους κινδύνους που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα αυτά παιδιά. Και βεβαίως και με συμμετοχή όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών, υπηρεσίες δικαιοσύνης, ε, κοινωνικές, κοινωνικών λειτουργών δηλαδή και ούτω καθεξής. Και θέλουμε να ανταλλάξουμε απόψεις με τις χώρες μέλη για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη συνεργασία αυτή. Με το δίκτυο δηλαδή για την ευαισθητοποίηση, τη ριζοσπαστικοποίηση RAN θα οργανώσουμε διάσκεψη αργότερα φέτος την Άνοιξη για τα παιδιά που επιστρέφουν. Με αυτό το θέμα δηλαδή. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εσείς λαμβάνετε πολύ σοβαρά υπόψη τα θέματα αυτά και μάλιστα αργότερα στην τρέχουσα εβδομάδα θα ε, συζητήσω με ορισμένου εξημών σε σχετική διάσκεψη για τα παιδιά που επιστρέφουν. Συζητούν επίσης οι εμπειρογνώμονες ε, και για τη δημιουργία δικτύων για την παρακολούθηση και είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε και να διευκολύνουμε την συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, εθνικών κυβερνήσεων δηλαδή, policy maker και τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και κάνουν την δουλειά αυτή στην οποία βασίζεται το RAN. Η ομάδα, η ομάδα αυτή συζητεί για την ενίσχυση των πρωτοβουλειών και ενεργειών και δραστηριοτήτων της Ένωσης και είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει και επίσης η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου θα συζητήσει και περαιτέρω μέσα στον χρόνο με ποιον τρόπο θα συνοδεύσει τις δραστηριότητες αυτές. Η ομάδα ασχολείται και με άλλα. Ιδεολογία, πόλωση, ριζοσπαστικοποίηση στην εξωτερική της διάσταση, επιγραμμική προπαγάνδα τι μπορεί να γίνει για την διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση και συμπερίληψη ή επανένταξη στην κοινωνία. Στις 9 Φεβρουαρίου οργανώνουμε συνάντηση με συμμετοχή των χωρών μελών για να προωθηθεί όλη αυτή η δουλειά και για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα εργασιών για το υπόλοιπο έτος. Ένα πιο συγκεκριμένο σημείο το οποίο θέλω να τονίσω, η έκθεση σημειώνει την ανάγκη να συνεχίσουμε την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας. Όπως γνωρίζουμε και από παλαιότερες συζητήσεις, το Ευρωπαϊκό Ιντερνετ Φόρουμ μας έχει επιτρέψει να συζητήσουμε με εταιρείε που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, με πλατφόρμες, για να μπορέσουμε κιόλα να προβάλλουμε αποτελεσματικά εναλλακτικά αφηγήματα στο διαδίκτυο. Αυτό έγινε και τον, και τον περασμένο Δεκέμβριο σε υπουργικό επίπεδο η συζήτηση αυτή. Αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να καλύψουμε. Στην τελευταία αυτή ανταλλαγή απόψεων τον Δεκέμβριο ζητήσαμε από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο να επιταχύνουν το, ε, την εργασία αυτή, δηλαδή στο κλείσιμο ιστοσελίδων με τρομοκρατικό περιεχόμενο, σε καλύτερη συνεργασία με τις Εθνικές Διοκτικές Αρχές και με την Ευρωπόλ, να συνεργαστούν καλύτερα οι μεγαλύτερες πλατφόρμες με τις μικρότερες, να υποστηρίξουν οι μεγαλύτερες τις μικρότερες, να εμποδίσουν το παράνομο αυτό περιεχόμενο να επανεμφανίζεται κάπου αλλού στο διαδίκτυο και ούτω καθεξής. Χρειαζόμαστε επίσης και εναρμονισμένη υποβολή ε, αναφορών, εκθέσεων για να μπορούμε να μετρούμε καλύτερα την πρόοδο στα διαφορετικά αυτά μέτωπα και στόχους. Για παράδειγμα, χρήση και αποτελέσματα της αυτόματης, αυτοματοποιημένης αναγνώρισης, ώστε να μην επαναφορτώνεται ένα σχετικό περιεχόμενο. Και πόσο αποτελεσματική είναι η προσπάθεια να εμπλακούν και οι μικρομεσαίες πλατφόρμες στην προσπάθεια αυτή. Οι συζητήσεις του Δεκεμβρίου για όλα αυτά τα θέματα αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμες. Ε, επί του παρόντος αξιολογούμε στο υποτοφός αυτών των συζητήσεων εάν και κατά πόσον χρειάζονται περαιτέρω βήματα για να εξασφαλιστεί περαιτέρω πρόοδος. Οι επιγραμμικές μας προσπάθειες βέβαια δεν περιορίζονται μόνο στην μείωση της τρομοκρατικής προπαγάνδας. Συμβάλλουν και στην προσπάθεια να τοποθετηθεί στο διαδίκτυο ένα καλύτερο αφήγημα. Εκεί χρειάζεται η συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να ανακοπεί η πορεία ορισμένων εκ των συμπολιτών μας προς μια ριζοσπαστικοποίηση. Ήδη από το 2016 έχουμε ξεκινήσει σχετικό πρόγραμμα με 10 εκατομμύρια ευρώ. Πέρσι το RAN με υποστήριξη ορισμένων από τους βασικότερους φορείς όπως Facebook, Google, Twitter βοήθησε πολλές πάνω από 200 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να εξετάσουν το είδος εκείνο ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για να μπορούν να προβάλλουν αυτό το θετικό αφήγημα. Ήδη έχουμε μια πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για ένα ποσό 60 εκατομμυρίων ευρώ που η σχετική πρόσκληση έκλεισε πριν από λίγες εβδομάδες και ελπίζουμε ότι θα δούμε ένα νέο κύκλο αυτού του νέου ε, αντιτρομοκρατικού αφηγήματος. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις πρακτικές για την προβολή αντιμηνυμάτων. Και αυτή η προσπάθεια είναι το ίδιο σημαντική και δύσκολη όπως και να αντιμετωπιστεί η δρομοκρατική προπαγάνδα στο διαδίκτυο γιατί είναι και δύσκολο να μετρηθεί η πρόοδος και η επιτυχία και της μιας και της άλλης ε, δυνατότητας, δηλαδή και της προβολής θετικών μηνυμάτων που θεωρούμε πάντως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβάλλονται δηλαδή εναλλακτικά αφηγήματα σε ομάδες στόχους. Παρόλες τις προκλήσεις αυτές ε, αρχίζουμε να βλέπουμε κάποια πρώτα θετικά αποτελέσματα οι, τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι stakeholders δηλαδή αρχίζουν να συνδυάζουν τις προσπάθειές τους εν τέλει ε, εκτιμώ ιδιαίτερα το ισχυρό θετικό μήνυμα Τη έκθεση, αντιλαμβανόμαστε ποιος είναι ο σημαντικός ρόλος του ΡΑΝ και άλλων σχετικών οργανισμών. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία, αναγνωρίζει το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και θα πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια στο δικό μας ευρωπαϊκό επίπεδο για να υποστηρίξει τις προσπάθειες των χωρών μελών, των αρχών των χωρών μελών και των νομικών επαγγελματιών στον χώρο αυτό, αλλά και αλλού, τον τομέα της ασφάλειας, ώστε να μπορέσει να επιτελεστεί σημαντική πρόοδο. Σας ευχαριστώ. Αυτό εδώ ολοκληρώνω την παρουσίασή μου. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις σε σχέση με την παρουσίασή σας, η κυρία Μετσόλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και εσάς, Επίτροπε Κίνγκ, που ήρθατε στην Επιτροπή μας Συμφωνούμε ότι τα κάτι μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης έχουν κάνει πολύ σπουδαίο έργο για να κρατήσουν ασφαλείς τους πολίτες μας. Έχουν περάσει πολλά νομοθετήματα και μετά τις επιθέσεις στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η εξέλιξη των γεγονότων δεν θα υποδαβλήσει μίσος και εχθροπρεξίες στις διαφορετικές κοινότητες που ζουν στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε να γίνει η Ευρώπη ένα έφορο έδαφο στρατολόγηση για του σκοπού των εξτρεμιστών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τρομοκράτε που είναι ε, υπήκοοι τη Ένωση, έχουν γεννηθεί εδώ, μεγάλωσαν στι κοινότητε τη Ευρώπη και ριζοσπαστικοποιήθηκαν ε, κατά την πορεία. Ε, θα θέλαμε λοιπόν μια πιο αυστηρή προσέγγιση για την καταπολέμηση τη ριζοσπαστικοποίηση, για την καταπολέμηση των εκφράσεων μίσου στι κοινότητέ μα και στο διαδίκτυο, να δούμε τι συμβαίνει στα σοφρονιστικά ιδρύματα, να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο των ξένων μαχητών και να δούμε τι ε, επιτρέπει στου ανθρώπου να γίνονται τόσο ευεπίφοροι στο να ριζοσπαστικοποιηθούν. Ε, όσον αφορά την επιγραμμική ριζοσπαστικοποίηση, συμφωνώ ότι η χρήση του ίντερνετ για σκοπούς τρομοκρατίας είναι κάτι που πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα ε, στο έργο μας. Πρέπει να εντοπίσουμε και να καταργήσουμε αυτά τα, αυτούς τους ιστοτόπους με τη διάδοση εκφράσεων και σκέψεων μίσους ε, ιδίως για τους πιο νέους, τους πιο ευάλωτους και για την καταπολέμηση των όσων ε, ισχυρίζονται οι τρομοκράτες στο διαδίκτυο. Δεν αρκεί απλώς να απομακρύνουμε το παράνομο περιεχόμενο, αλλά να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν και τις συνέπειες ε, του να υπάρχουν ε, πληροφορίες ε, για το τι πραγματικά επιδιώκει η προπαγάνδα με αληθινές εικόνες το τι προκαλεί η ριζοπαστικοποίηση. Πρέπει να συνεργαστούμε με όσους είναι φορείς του διαδικτύου, εταιρείε και ενδιαφερομένους και όλες τις αρμόδιες ομάδες. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το δίκτυο για την ευαισθητοποίηση στη ριζοπαστικοποίηση και τον είπα το Επίτροπο για το θέμα αυτό και θα πρέπει να φροντίσουμε η έλλειψη ελπίδα και προοπτική για τους νέους και τι κοινότητές μας να μην μεταφράζεται στο ότι ο εκτρεμισμό, οι ακραίε τάσεις είναι η μόνη διέξοδος και ότι η έλλειψη ελπίδα εκπαίδευση του κάνει εύκολη λία για, την, ε, για του σκοπού τη τρομοκρατία. Πρέπει να το ε, καταγράψουμε. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα συμπεράσματα να τεθούν σε εφαρμογή, να, να συνεργαστούμε καλύτερα για τις συστάσεις και να δούμε ποιοι, ποιες άλλες λύσεις μπορούμε να σκεφτούμε σε επίπεδο ένωσης, πέραν των όσων ήδη έχουμε για να καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση. Ευχαριστούμε κυρία Σίπελ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για αυτή σας την ε, εισήγηση. Να τονίσω ότι όταν μιλάμε για ριζοσπαστικοποίηση σε ισοφρονιστικά ιδρύματα, σε καταπλησμούς προσφύγων, μια σχετική μελέτη την κάναμε και στη Γερμανία για το σκοπό αυτό, για το ρόλο των θρησκευτικών ηγετών, πρέπει να βρούμε τρόπους ε, να αναπτύξουμε αντίρροπες δυνάμεις. Συμφωνούμε όλοι. Όμως, για την όλη εξέλιξη της ένταξης. Να πω ότι μερικοί ριζοσπαστοκοποιούνται επειδή ίσω δεν αισθάνονται για αίσθημα της κοινωνίας, δεν έχουν εκπαίδευση, δεν έχουν ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση. Αλλά δεν είναι πάντοτε μόνο αυτή η αλήθεια. Κάποιοι όχι απλώς γεννήθηκαν σε κάποια από τα κατημέλη μέλη μας, αλλά και οι γονείς τους έχουν γεννηθεί σε κάποια από τα κράτη-μέλη μας και έχουν διαβατήριο ενός από τα κράτου, κράτη-μέλη μας. Όμως, ακόμα θεωρούνται ξένοι. Θα δώσω το παράδειγμα κάποιου που οι γονεί του γεννήθηκαν εδώ, που κατοικεί εδώ, έχει γερμανικό διαβατήριο και το ρωτήσανε για πες τι άποψη έχεις για τις τελευταίες δράσεις του Πρόεδρου και είπε «Στάνμαγερ». Αυτόν εννοείς. Όχι, τον δικό σου Πρόεδρο. Τον Ερντογάν. Ε, αυτό συμβαίνει, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ζουν στις κοινωνίες μας και ακόμη και με καλά προσόντα μπορεί να μην αισθάνονται μέρος της κοινωνίας και κινδυνεύουν να τους προσελκύσουν άνθρωποι που προσπαθούν να οδηγήσουν άλλους στον εξτρεμισμό. Όταν μιλάμε για παιδιά, παιδιά που ανατράφηκαν στη Συρία, την Γερμανία ή άλλες χώρες, πρέπει να σκεφτούμε τι συμβαίνει. Απλώς μεγάλωσαν σε εξτρεμιστικά περιβάλλοντα ή εκπαιδεύτηκαν να είναι εξτρεμιστές οι ίδιοι και να δράσουν ως τρομοκράτες. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη θεώρησή τους για τη ζωή. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τους οικογενειακούς τους δεσμούς και τις οικογένειές τους. Έχουμε κάποιες ανταλλαγές απόψεων με άλλες χώρες όπου βρίσκουμε παιδιά να έχουν ήδη στρατιωτική δράση Μπορούμε λοιπόν ίσως να υποφεληθούμε από, τη δική τους την, ε, από το δικό τους παράδειγμα, τη δική τους εμπειρία. Και κάτι άλλο που θέλω να τονίσω είναι ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε για ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ένας από τους υπο, ένα από τα υποκείμενα αίτια ε, πολέμου και επιθέσεων από τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τρόπος ακριβώς που μεταχειριζόμαστε τις τρίτες χώρες έχετε καμία συνεννόηση στη δική σας υπηρεσία με τις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης της Επιτροπής και των κατών μελών για να δείτε πώς η δική μας προσέγγιση για την ενίσχυση της δημοκρατίας, της ειρήνης και της πραγματικές εταιρικές σχέσεις με άλλες χώρες μπορεί μακροπρόθεσμα τελικά να γίνουν ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση. Ευχαριστούμε κυρία Στίβενς για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Κιν για την παρουσίασή του. Είναι σημαντική δουλειά την οποία έχει κάνει μέχρι τώρα. Μία από τις ερωτήσεις μου είναι το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει και να συνδράμει τις εταιρείες των κοινωνικών μέσων δικτύωσης όπως το Twitter και να τις καταστήσει ικανές να βοηθήσουν στον αγώνα των δικό μας εναντίον της ροζοσπαστικοποίησης. Νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε και να παρακολουθούμε τα δικαιώματα και τον σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης και ταυτόχρονα είναι δύσκολη βέβαια η ισορροπία αυτή, αλλά σας στηρίζω στην προσπάθεια την οποία κάνετε εναντίον της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης. Γνωρίζω ότι στο στις Ηνωμένε Πολιτείες το Κογκρέσο αποφάσισε να ακολουθήσει τη λεγόμενη εκ του μακρόφεν αντιμετώπιση, hands off αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις ακολουθούν τις δικές τους μεθόδους και μέσα. Εμείς νομίζω ότι πρέπει να εμπλακούμε στην συζήτηση αυτή και δεν μπορούμε να αφήσουμε ελεύθερες και μόνες τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν την υπόθεση αυτή. Περαιτέρω, έχετε την δυνατότητα να μας παρουσιάσετε μια επισκόπηση των χρηστών πρακτικών στις διάφορες χώρες στον τομέα της απορριζοσπαστικοποίησης. Ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία έχουμε είναι ότι οι ιδέες έχουμε πολλές και καλές. Κάποιες όμως δεν είναι λειτουργικές. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί έτσι ώστε οι χρηστές αυτές πρακτικές να διαδοθούν όπως πρέπει. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρονται στις ε, στρατηγικές αυτές των που ακολουθούν οι επιχειρήσεις ε, στο διαδίκτυο για να μας δώσουν την εξήγηση ε, για το είδος του αφηγήματος, του αντιαφηγήματος το οποίο αυτές προτείνουν. Έτσι θα μπορέσει ίσως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει το πού βρίσκεται σήμερα. Η κυρία Βίξτρομ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τον Επίτροπο που ε, ήρθε να μας επισκεφτεί Ευχαριστώ επίσης και για τις λεπτομερέστατες απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις μου τις γραπτές πρόσφατα. Είναι σαφές ότι πρέπει όλοι να εμπλακούμε στη συζήτηση αυτή και όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε λίγο για το λεγόμενο αντιαφήγημα για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίηση. Και θα ήθελα να επανέλθω και στην ερώτηση για την ριζοσπαστικοποίηση ε, σαν κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο οριζών. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στα κράτη-μέλη, τα οποία θα πρέπει να ανταμοιραστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε όχι μόνο να επενδύσουμε μόνο χρόνο και ενέργεια, επανεφευρίσκοντας ε, τον τροχό επανειλημμένα. Νομίζω ότι μια από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις είναι ότι άκουσα εδώ στο Βέλγιο μία περίπτωση όπου έχουν ε, μάλλον προσλαμβάνονται ουσιαστικά, στρατεύονται, ακούγεται ε, από πάρα πολλές κοινότητες ε, παιδιά στον Ισλαμικό στρατό, ενώ η δουλειά που έχει γίνει σε πολλές περιοχές από αυτές που θεωρεί το δεδομένο ότι υπάρχει στράτευση προς το Ισλαμικό κράτος, κάτι τέτοιο δεν ισχύει πλέον, λόγω επαναλαμβάνω της καλής δουλειάς που έχει γίνει. Ταυτόχρονα μιλάμε για το τι συμβαίνει στο διαδίκτυο σαν να είναι κάτι το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι παράνομο στην πραγματικότητα είναι παράνομο και διαδικτυακά. Εμείς ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά είχαμε συζητήσει τα θέματα αυτά των παράνομων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο και νομίζω ότι η πραγματική ζωή και το διαδίκτυο δεν διαφέρουν ιδιαίτερα και όταν υπάρχουν επινικές κολάσιμα ποινικά ε, ε, ενέργειες στην πραγματική ζωή πρέπει αντίστοιχα να ε, Ισχύει το ίδιο και για το διαδίκτυο. Τώρα για την αντιμετώπιση των, των λόγων και των αιτιών που δημιουργούν την ριζοσπαστικοποίηση σε βάθος της τρίτες χώρες. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα αν θέλουμε κάτι να επηρεάσουμε. Πάντως σας ευχαριστώ για μια ιδιαίτερα πλήρη παρουσίαση. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εξετίμησα το ότι ήρθατε πάλι εδώ μαζί μας σήμερα και μας μεταφέρατε ένα σαφές μήνυμα. Η ερώτησή μου, όπως πολύ σωστά είπατε, ο ρόλος της θρησκείας και των θρησκευτικών ηγετών, ιδιαίτερα όταν είναι φυλακισμένοι, είναι κάτι το οποίο σε πάρα πολλές περιπτώσεις οδηγεί στην εκκίνηση, αν θέλετε, της ε, ριζοσπαστικοποίησης σε βάθος. Ε, είναι κάτι το οποίο διαφεύγει της προσοχής των τοπικών αρχών, των αρχών γενικά. Και εδώ οι τοπικές αρχές, σαν παράδειγμα, και γνωρίζω ότι και από τη δική μου χώρα, έχουν αρχίσει να αναζητούν χρηματοδότηση από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία για να χρηματοδοτήσουν ετεμένη και κοινωνικές Ισλαμικές δομές. Αυτό στην αρχή ακούγεται σαν κάτι το αρκετά ευχάριστο και εύκολο, χωρίς να γνωρίζουν τις επιπτώσεις. Ε, υπάρχει λοιπόν συνειδητοποίηση σταδιακά στα διάφορα κράτη-μέλη για το αρνητικό αυτή της αντιμετώπισης. Ποια είναι τώρα η άποψή σας μετά από τις προπαρασκευαστικές ε, ε, εκθέσεις γενικά γύρω από το θέμα των ε, διαχωρισμένων πληθυσμών στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Ξέρουμε ότι οι φυλακές λειτουργούν σαν κέντρα ριζοσπαστικοποίησης, οπότε κάποιοι πιστεύουν ότι απομονώνοντας και ξεχωρίζοντας αυτούς οι οποίοι παρουσιάζουν υποτίθεται υψηλούς κινδύνους εξτρεμιστικών και ακραίων ιδεών, Κάτι τέτοιο ε, θα διευκολύνει την μη επιμόλυνση των υπολείπων. Δυστυχώς όμως από ό,τι φαίνεται δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι για λόγους αποκατάστασης, διόρθωσης της πορείας τους και κατανόησης αυτών τα οποία θεωρούν κάτι τέτοιο είναι λάθος. Τώρα, τι πιστεύετε για τα κράτη-μέλη που πιστεύουν ότι θα επιτρέψουν σε Ευρωπαίους πολίτες ε, να δικάζονται σε τρίτες χώρες. Σε τρίτες χώρες οι οποίες θα έλεγα δεν έχουν και ιδιαίτερα μεγάλη φήμη για τα δικαστικά του συστήματα όπως το Ιράκ, η Συρία κτλ. Αν επιτρέψουμε στους ανθρώπους αυτούς ε, να δικαστούν σε αυτές τις χώρες είναι σαφές ότι δεν θα δικαστούν ουσιαστικά ή η δίκαιη δίκη στην οποία έχουν δικαίωμα δεν θα υπάρχει. Συνεπώς λοιπόν θέλω και εδώ την άποψή σας. Λοιπόν, επιγραμμική αντιμετώπιση και αντίθεση στα τρομοκρατικά μηνύματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει με σωστά μηνύματα. Καταρχάς απαιτούνται εμπειρογνώμονες σε επίπεδο γλωσσικό. Χρειαζόμαστε εμπειρογνώμονες του Ισλάμ για να μπορέσουν να δώσουν το σωστό μήνυμα και να μην λειτουργήσει κάτι τέτοιο αντιπαραγωγικά. Σε ποιο βαθμό εσείς πιστεύετε ότι αυτό ανήκει στους ρόλους τους οποίους πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ποιο βαθμό στα κράτη-μέλη. Τέλος, πρόσφατα έμαθα ότι η δουλειά την οποία κάνουν οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών μηνυμάτων είναι ελάχιστη ουσιαστικά. όχι μόνο για τους ε, τζιχαντιστές αλλά και για τους ακροδεξιούς οι οποίοι πολλές φορές δυστυχώς ε, πολλαπλασιάζονται στην επιγραμμική ε, παρουσία τους. Εγώ δεν έχω διαπιστώσει αδίποτε μορφή δράσης γύρω από τα θέματα αυτά και υπάρχουν πάρα πολλοί επικίνδυνοι άνθρωποι της άκρας δεξιάς στο διαδίκτυο. Κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, Επίτροπε, ε, για την παρουσίαση εδώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Κατά πρώτον, συμφωνώ ότι οι φυλακές, τα σοφρονιστικά ιδρύματα, είναι ακριβώς μερικά από τα σημεία όπου κατεξοχήν μπορεί να πέσουν θύματα στρατολόγησης, ριζοσπαστικοποίησης ε, οι φυλακισμένοι, ιδίω εφόσον είναι μουσουλμάνοι. Όμως δεν είναι μόνο οι φυλακές. Γι' αυτό έχω μια-δυο ερωτήσεις. Κατά πρώτον, έχετε καμία ιδέα τι συμβαίνει στα τζαμιά, τα τεμένη των ε, μουσουλμάνων τι συμβαίνει με τα κηρύγματα που εκφωνούνται εκεί, ε, ποια είναι η δράση που καλλιεργείται, ποιε οι κουβέντε που γίνονται. Και επίση ω προ την καταπολέμηση τη ριζοσπαστικοποίηση. Μιλήσατε με θρησκευτικού ηγέτε των μουσουλμανικών κοινοτήτων στα κράτη-μέλη Πιστεύετε ότι αν δεν είναι με το πλευρό μας μπορούμε να τα καταφέρουμε, πρέπει να τους πείσουμε ότι ε, έχουμε έναν κοινό αγώνα για να καταπολεμήσουμε την ριζοπλαστικοποίηση. Ευχαριστούμε κυρία Ντεπρέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο Κίνγκ και γιατί έρχεται πολύ συχνά στην Επιτροπή μας και μας ενημερώνει, αλλά και ό,τι μας λέει είναι και πολύ ξεκάθαρο και σαφές. Έχω δύο ερωτήσει Επιτροπέ, διάβασα την ενδιάμεση έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου για την σοσπαστικοποίηση και βρήκα καλές συστάσεις που θα πρέπει βεβαίω να μελετηθούν περαιτέρω, να δούμε τις καλές πρακτικές και ούτω καθεξής. Ε, αναγκαίο αυτό, αλλά κάτι άλλο μου φαίνεται πιο θεμελιώδες. Θα έρθουν διάφοροι... Τρομοκράτε από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μπορεί και να μην επιστρέψουν, διότι τα διάφορα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικέ πολιτικέ ω προ του τρομοκράτε που έχουν πάει στη Συρία και το Ιράκ και ε, τα διάφορα παιδιά επίση. Δεν θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να εναρμονίσουν του κανόνε του προ το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα για το καθένα από τα κράτη-μέλη. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ε, εκατοντάδα παιδιά θα ξανάρθουν για την ώρα θα προσπαθήσουμε να του ενσωματώσουμε. Σε λίγα χρόνια θα ενηλικιωθούν. Εάν ριζοσπαστικοποιηθούν, πώ θα αντιδράσουμε. Μόνο η χώρα που θα του υποδεχθεί θα είναι ε, υπεύθυνη. είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, το καταλαβαίνω, αλλά τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να προσπαθήσουν να αναρμονίσουν τη στάση του. Και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων, δεν το συζητώ αυτό καν. Ε, αλλά κάτι το κοινό θα έπρεπε να γίνει λογικά πέραν από την ανταλλαγή δεδομένων. Ε, κυρία Σίπελ, θα συμφωνήσω ότι υπάρχει μια κοινωνική διάσταση στην ε, πρόκληση της ριζοπαστικοποίηση. αλλά όχι μόνο αυτό. Κάποια, ε, ο, κάποιος από την υπηρεσία της Επιτροπής ο κύριος Σάρντ Αντραμέ που είναι Βέλγος, μαροκινής καταγωγή και ειδικευμένο στα θέματα της ε, καταπολέμησης τη βασιλικοποίησης μα είπε ότι υπάρχουν και άλλες διαστάσεις πέραν της αστυνομικής καταπολέμησης. Ε, πρέπει να δούμε την καταπολέμηση όχι μόνο στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να δούμε τα θεμέλια, τη γενεσιουργικά αίτια των όσων τροφοδητούν την ζωοφροντικοποίηση. Α πούμε, ας δούμε, ας πούμε, την, ε, το δρόμο του Μαρόκου. Ένα Ινστιτούτο για την εκπαίδευση των ημάμιδων και η απαγόρευση της δημοσίευσης ε, βιβλίων ε, με ριζοσπαστική ας πούμε διάσταση είναι κάτι που συνέβη στη χώρα. Δύο μέτρα που έλαβε η χώρα αυτή. Δεν πρέπει να απευθυνθεί λοιπόν μια έκκληση στις θρησκευτικέ αρχές ώστε ακόμα και η ίδια εκπαίδευση των ημάμιδων να γίνει με άλλο τρόπο, με άλλη διαδικασία από αυτήν την πολεμοχαρή και ζωοπρακτικοποιημένη που έχει επικρατήσει. Λογικό είναι οι πολιτικέ αρχέ να προσκαλέσουν άλλε αρχέ με επίση μεγάλο κύρο και βαρύτητα να λάβουν μέτρα για να καταργηθεί μία από τι ρίζε, ένα από τα γενεσιουργά αίτια τη ροσπαστικοποίηση, εφόσον γίνεται. Εκεί ήθελα την άποψή σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κιέγκε. Ευχαριστώ. Κλοντ, ευχαριστώ Επίτροπε για όσα έχετε κάνει και όσα μας παρουσιάσατε γνωρίζουμε ότι η καταπολέμηση κάθε μορφής ρίζοσπαστικοποίησης και ε, βίαιου εξτρεμισμού απαιτεί ε, μια πανοπλία μέτρων από την πρόληψη ως την εκπαίδευση και επίσης μέτρα που θεωρούνται και κατασταλτικά σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα κάποιες φορές. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τις πολιτικές ένταξεις. Ήδη μιλήσαμε για αυτές. Βλέπουμε ότι σε πολλές χώρες η διάσταση αυτή έχει πολλές ελλείψεις. Να ξεκινήσω με κάποιες πτυχές που κατά την άποψή μου πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ε, οπτική του να εναρμονίσουμε κάποιους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπηκότητα. Πολλά από τα παιδιά αυτά δεν αισθάνονται ότι ανήκουν σε κάποιο κράτος από τη μια, γιατί η αναγνώρισή τους στην επικράτεια δεν τους δίνει καθεστώς που να επιτρέπει από όταν είναι μικρά να θεωρήσουν ότι ανήκουν σε μια συγκεκριμένη επικρατεία και περιμένουν 18-20 χρόνια για να αναγνωριστεί ότι είναι παιδιά ενός κράτους. Είναι παιδιά που βρίσκονται σε ένα λίμπο, σε μια ενδιάμεση κατάσταση, χωρίς να έχουν ίσες ευκαιρίες όπως οι συνομιλικοί τους της ίδιας χώρας. Αυτό θα ήταν ένα σημείο επί το οποίο θα μπορούσαμε να αναλάβουμε δράση. Ακόμη και η ομάδα ε, ψηλού επίπεδου θα μπορούσε να το σκεφτεί και να το μελετήσει για να οδεύσουμε προς μία εναρμόνιση. Δεύτερη παρατήρηση σε ό,τι αφορά την αύξηση του μίσους, την ένταση του μίσους, ε, του λαϊκισμού και της ξενοφοβίας. Δεν πιστεύετε ότι στον κόσμο αυτό μια τόσο ε, τιμωρητική προσοχή που δίνεται ιδίω για να ελέγξουμε την εξάπλωση του μίσους σε μια χώρα δεν ε, βάζει σε, δεύτερο, σε δεύτερη μοίρα ακόμα και τις πολιτικές της πρόληψης. Διότι όσο πιο πολύ υπάρχει αντιπαράθεση προς κάποιες κοινότητες μέσα σε μια χώρα, πιο δύσκολο είναι να υλοποιήσει κανείς πολιτικές πρόληψης. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, εάν από τη δική σας την οπτική γωνία σκεφτήκατε καθόλου και αυτήν τη διόγκωση των φαινομένων όπως το μίσος και η ξενοφοβία, που μπορεί να αποτελέσουν ε, φραγμό για να σχεδιαστούν και καλές πολιτικές πρόληψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντεχόφσκι. Ευχαριστώ. Επίτροπε, ευχαριστούμε που ήρθατε και παρόλο που είναι Δευτέρα απόγευμα, εμείς πάντοτε ερχόμαστε στις ακροάσεις σας και ακούμε τι έχετε να μας πείτε. Χαίρομαι πολύ που είπε όσα είπε η κυρία Σίπελ, διότι είναι η πρώτη φορά που έκανε μια τόσο λογική ανάλυση της μεταναστευτικής κρίσης και της ανάγκης να ενταχθούν οι πολίτες που έρχονται στην Ευρώπη, διότι στο παρελθόν είχα ακούσει απόψεις όπως θα πρέπει να δεχόμαστε και να καλωσορίζουμε τους πάντες και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, θέλω να τονίσω το θέμα της ένταξης. Συμφωνώ απολύτως με την κυρία Σίπελ. Ε, μη μου ξαναπείτε όμως ότι το ΕΛΚ δεν μπορεί να συμφωνήσει ποτέ με τους σοσιαλιστές. Δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, τα αφήνω αυτά και θέλω να ρωτήσω τρία πράγματα. Πρώτον, ριζοσπαστικοποίηση μέσω ψευδών ειδήσεων. Ε, ακόμη και εγώ ο ίδιος και η οικογένειά μου ε, λάβαμε απειλές ε, για δολοφονία ε, λόγω των ψευδών ειδήσεων. Πώς το αναχαιτίζεται αυτό το φαινόμενο. Διότι ο κύριο Ντράχος, ο, πρόεδρος, ε, ο υποψήφιος πρόεδρος στην προεκλογική εκστατεία για τι προεδρικές εκλογέ τη Τσεχίας, επίση με ψευδείς ειδήσει βρέθηκε να λέει ότι θέλει να καλωσορίσει μετανάστε στη χώρα μα και δέχτηκε απειλέ για τη ζωή του. Δεύτερο ερώτημα ε, για την ριζοσπαστικοποίηση μέσω τη ρωσική προπαγάνδα. Ένα θέμα που συζητιέται πολύ στη δημοκρατία τη Τσεχίας. Ένα θέμα που είναι πολύ ε, καυτό, διότι είναι πολύ έντονη η προπαγάνδα των ρωσικών μέσων ενημέρωσης και προκαλεί τη ριζοπαστικοποίηση κάποιων. Και τρίτον, για κάποιες περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού. Εγώ εργάστηκα ως υπάλληλο των δημοτικών αρχών στις κινητές υπηρεσίες για πολλά χρόνια και βλέπω ότι η έλλειψη κινητικότητας καλλιεργεί φαινόμενο όπως η ζωσπαστικοποίηση. Ισχύει σε πολλές χώρες. Είναι κάτι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να σκεφτούμε στο μέλλον. Δεν ξέρω αν έχει άμεση σχέση με το θέμα, Τόμας, αλλά θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει σε αυτή και πολλές άλλες ερωτήσεις εφόσον θέλει. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ όλους που ασχολείστε με τα θέματα αυτά. Είναι σημαντικά θέματα και πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί προετοιμάζοντας την επόμενη φάση των εργασιών των εμπειρογνωμόνων. Επαναλαμβάνω ότι η έκθεση αυτή είναι ενδιάμεση και θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω κάποιες ερωτήσεις που προέρχονται συνήθως από διαφορετικές κατευθύνσεις Τώρα η πρόκληση την οποία δημιουργεί η επιγραμμική προπαγανδιστική τρομοκρατική δραστηριότητα. Εμείς όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια δημιουργούσαμε, δημιουργήσαμε διάφορες πλατφόρμες συζήτησης των θεμάτων αυτών με τους εκπροσώπους της διαδικτυακής βιομηχανίας και τα κράτη-μέλη. Η κυρία Γιούροβα, σαν παράδειγμα, έχει συμφωνήσει ένα κώδικα συμπεριφοράς ε, για, το, για την ρητορική μίσους. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει ασχοληθεί με το περιεχόμενο στα φόρα του ίντερνετ της τρομοκρατίας και ο κύριος Σάνσιπ και Γκάμπριελ μέχρι πιο πρόσφατα ε, έχει ασχοληθεί με διάφορες πλατφόρμες έτσι ώστε ε, να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο τεχνολογικό στο διαδίκτυο η ρητορική του μίσους και της τρομοκρατίας. Προσπαθήσαμε λοιπόν από πέρυσι να συντονίσουμε τις μορφές αυτού διαλόγου και να καταλήξουμε σε κάποια ενιαία, αν θέλετε, πρακτικά βήματα Γι' αυτό οδηγηθήκαμε το Σεπτέμβριο του 2017 σε μια νέα ανακοίνωση, ελπίζω να μπορέσατε να τη διαβάσετε, που ξεκαθαρίζει ακριβώς το τι επιτρέπεται στο διαδίκτυο και το τι μπορεί να γίνει στο διαδίκτυο για να αντιμετωπιστεί το παράνομο περιεχόμενο διαφορετικής προέλευσης. Και προσπάθησαν να διευκρινίσουν ότι υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν να γίνουν και οφείλουν να γίνουν έτσι ώστε να λειτουργήσουμε προληπτικά και σε επίπεδο αυτοματοποιημένο να εντοπίζουμε και να κλείνουμε και να απαγορεύουμε και τη φόρτωση τέτοιου είδους περιεχομένου. Και θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να επηρεάσουμε αρνητικά το πλαίσιο το νομικό ανάληψη ευθύνης ε, των εμπορικών συναλλαγών στο διαδίκτυο. Συνεχίζουμε λοιπόν να δημοσιεύουμε εκθέσεις ε, στα πλαίσια αυτών των διαλόγων και επαφών. Η κυρία Γιούροβα της πριν δέκα μέρες δημοσίευσε κάποια σημαντικά στοιχεία προόδου θα έλεγα για την προληπτική αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Αναφέρθηκα επίσης και στη συνάντηση για το διαδίκτυο που έγινε τον Δεκέμβριο. Έγινε λοιπόν κάτι, έχουμε προχωρήσει κάπως, υπάρχουν βήματα προόδου, μένει να γίνουν περισσότερα σε σχέση με τις παράνομες τρομοκρατικές ε, δραστηριότητες Εκεί θα έπρεπε ε, να ε, βελτιωθεί η ταχύτητα ταυτοποίησής τους και κλεισίματός τους, να χρησιμοποιηθούν ακόμα περισσότερο αυτοματοποιημένα συστήματα έτσι ώστε να μην φορτώνονται τα sites αυτά και θέλουμε επίσης ε, να μπορέσουμε να ασχολούμαστε όχι μόνο με τις μεγάλες πλατφόρμες αλλά και με τις νεοπαγείς επιχειρήσεις του διαδικτύου, τις νέες πλατφόρμες μικρού μεγέθους και θα θέλαμε λοιπόν να υπάρξει και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους σερβερς αυτούς και τις αρχές τις κατασταλτικές σε επίπεδο ευρωπαϊκό και εθνικό. Υπάρχει συνεργασία, μένει να βελτιωθεί. Αυτή είναι λοιπόν η βασική μας δραστηριότητα τώρα. Στην Επιτροπή αυτή την εποχή συζητάμε για το πώς θα μπορέσουμε εμείς να ενθαρρύνουμε αυτού του είδους την πρόοδο, για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τις προσπάθειές μας αυτές να καρποφορήσουν είτε το Φεβρουάριο είτε αμέσως μετά. Νομίζω λοιπόν ότι μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το θέμα αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη και προσπαθούμε να το προχωρήσουμε με συντονισμένο τρόπο. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ερωτήσεις τις οποίες δεν μπορώ να απαντήσω λεπτομερώς, θα απαντήσω όμως κάπως γενικά. Υπάρχει καταρχάς πάρα πολλή δουλειά η οποία γίνεται σε σχέση με, τους, με, τους, με τα παιδιά τα οποία επιστρέφουν. Νομίζω ότι έχει συνταχθεί ένα, στα μέσα του 17 ένα πολύ σωστό εγχειρίδιο, χρήσιμο εγχειρίδιο που προκάλεσε αρκετές συζητήσεις στα κράτη-μέλη. Υπήρξαν επίσης και ανταλλαγές που διευκολύθηκαν από το ΡΑΝ και σε υπουργικό επίπεδο για τις προκλήσεις που θέτουν οι ξένοι μαχητές, ε, της ενημέρωσης αν το πράγματι επιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς ελέγχονται από το δικαστικό σύστημα. Είναι βασικό θέμα το οποίο ε, συζητιέται στα ε, προγεύματα εργασίας τα οποία οργανώνει το Υπουργικό Συμβούλιο ε, και επίσης το τι γίνεται σε επίπεδο εθνικό. Το θέμα σαν παράδειγμα του διαχωρισμού στις φυλακές, όπου κάθε χώρα έχει τις δικές της πρακτικές. Το τι θέση λαμβάνει καλής σε σχέση με τις ε, δικαστικές ε, αντιμετωπίσεις στους τρίτες χώρες. Κάθε χώρα και εδώ λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά θα μας βοηθήσουν ε, ε, στο να καταλήξουμε κάπου έτσι ώστε να περιλαμβάνονται και στην επόμενη έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Τώρα για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, για την πρόκληση την οποία παρουσιάζει η συνεργασία με τις τρίτες χώρες και σε ποιο βαθμό ενθαρρύνουν την ριζοσπαστικοποίηση. Να κάνω τη διάκριση εδώ ε, ανάμεσα στις γενικές επιρροές που μπορεί να έχει η εξωτερική μας πολιτική, σαν παράδειγμα η ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή, Αυτά είναι θέματα τα οποία συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η ειδικού τύπου προκλήσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες εταίρους για την αντιμετώπιση της ζωσπαστικοποίησης στις χώρες αυτές και σε ποιο βαθμό μπορούμε να επηρεάσουμε αυτούς τους ε, ριζοσπάστες οι οποίοι διαδίδουν τα μηνύματά τους και εκεί και εδώ και τι μπορούμε να κάνουμε στη συνεργασία και στην ενθάρρυνση με τον δε. Αυτά λοιπόν συζητιώνται στα πλαίσια των διαλόγων ε, σε θέματα ασφαλείας ε, με όλους τους γείτονες και εταίρους. Τώρα για τα θέματα της ολοκλήρωσης ενσωμάτωσης. Εμείς αναγνωρίζουμε και πολλοί από εσά το είπαν από διαφορετικές προοπτικές ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του εύρους των πολιτικών τα οποία είναι στη διάθεσή μας στον τομέα αυτό. Υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης ένταξης το οποίο εξελίσσεται εδώ και αρκετά χρόνια και ταυτόχρονα ε, πριν από λίγο καιρό η Επιτροπή δημοσίευσε μια εργαλειοθήκη η οποία βοηθά τις χώρες να χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα διαθέσιμα ταμεία της Ένωσης για να βοηθήσουν την ένταξη των μεταναστών, των νεοαφιχθέντων μεταναστών. Λοιπόν, αυτό αναφέρεται στην παρούσα χρηματοδοτική περίοδο μέχρι το 20. Θέλω να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω εδώ τις εργασίες ε, της Αρμόδιας Επιτρόπου. Τώρα, στο τι μαθήματα μπορούμε να έχουμε πάρει από τα κράτη-μέλη γύρω από τα θέματα αυτά και ποιες είναι οι χρηστές πρακτικές. Μα αυτός είναι ο στόχος αυτής της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου. Ελπίζω ότι όταν επανέλθουμε τελικά με κάποιες προτάσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας να μπορέσουμε επιτέλους να κάνουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες να ισορροπούν ανάμεσα στο τι μαθαίνουμε από αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο φυλακές αλλά εκπαίδευση, κοινωνική, λειτουργή, και άλλα θέματα που έχουν σχέση με τις συνέπειες της ριζοσπαστικοποίησης και από την άλλη αυτούς που χαράσουν τις πολιτικές στις διάφορες χώρες. Αυτός είναι ο σύνδεσμος τον οποίο εμείς θέλουμε να αποτελέσουμε και αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα της επόμενης φάσης εργασιών της ομάδας υψηλού επίπεδου. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος Μωράης, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε καθώς και τις και τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις τους βεβαίως. Πρόκειται για την πραγματική τομή ε, του θέματος και για τις νομοθετικές πρωτοβολίες βέβαια. Ευχαριστώ και για την συνεργασία των επιτρόπων μεταξύ τους. Θα σας προσκαλέσουμε και πάλι όταν θα εκδοθεί η νέα έκθεση της ε, ε, Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για ε, εμπειρογνωμόνων, μάλλον, ομάδας εργασία, εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου. Όταν θα έχουμε την επόμενη έκθεση, λοιπόν, θα σα προσκαλέσουμε και πάλι, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, να προχωρήσουμε τώρα αμέσω στο επόμενο θέμα τη ημερησία διατάξεως, που είναι η πρόεδρος της ομάδας εργασίας άρθρου 29, την οποία παρακαλώ να προσέλθει στα έδρανα του Προεδρείου. η, ε, πρώτη την κυρία Ισαμπέλ Φάλκε Πιερωτά, η οποία θα μας παρουσιάσει την έκθεση για την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Θα θυμάστε ότι η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 συμμετέσχε στην πρώτη ε, αυτή, ε, έχει μάλλον κάνει μια πρώτη έκθεση και θα μας μιλήσει η κυρία Πιερωτά για το έργο της ομάδας εργασίας του άρθρου 29. Ε, θα ήθελα να θυμίσω ακόμη ότι είχατε μια εξαιρετική θητεία ε, και σε άλλες θέσεις και ιδίως για τις ορισμένες δραστηριότητες που έχετε αναλάβει σας ευχαριστώ για αυτές, αγαπητή Ισαμπέλ, και σας παρακαλώ να προβείτε στην παρουσίασή σας. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Σας ε, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας απευθύνω το λόγο για δύο θέματα πραγματικά σημαντικά. Αφενός την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και αφετέρου τη ΓΚΠΔ. Και ευχαριστώ για τα όσα είπατε για την Προεδρία του άρθρου 29. Πρώτα, για την ασπίδα προστασία της ιδιωτική ζωής. Πώς γνωρίζετε το άρθρο 29 που άρχισε το προηγούμενο, ε, το προηγούμενο έτος έχει γίνει τώρα βέβαια έγκριση της νέας αυτής προτάσεως για τη μεταφορά ε, προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ. Στόχος της επανεξέτασης αυτής για τις αρχές προστασίας δεδομένων ήταν διπλός. Αφενός ε, να διαβεβαιωθούμε ότι οι αμερικανικές δεσμεύσεις για την προστασία της αδειωτικής ζωής πραγματιτηρούνται και δεύτερο για να συνεχίσουμε την ανάλυση που είχε ήδη αρχίσει στη γνωμοδότηση του Ιουλίου 2016 για την συμβατότητα με το δίκαιο των συνθήκων αλλά και το δευτερογενές δίκαιο των ευρωπαϊκών ε, συνθήκων δηλαδή ε, και για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίναμε έκθεση τον Νοέμβριο 2017, στην οποία έκθεση αναγνωρίζουμε τις προόδους που έχουν γίνει σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις που προσφέρει ε, η ασπίδα προστασίας ιδιωτικής ζωής σε σχέση με τον ασφαλή λιμένα και βεβαίως τις δεσμεύσεις που υλοποιούν οι Αμερικανοί. Και πρώτα για ζητήματα εμπορικά. Μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ενίσχυση ελέγχων και παληθεύσεων πριν από την εγγραφή στο μηχανισμό των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Από την άλλη μεριά, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και οι αυτόματες διαδικασίες πρέπει ακόμη να βελτιωθούν. Τέλος, το άρθρο 29 σημειώνει την έλλειψη ρυθμίσεων για ορισμένα πρόσωπα όταν τα προσωπικά τους δεδομένα μεταφέρονται για λόγους εμπορικούς στις ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά τα σχετικά με την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από τις Αμερικανικές Αρχές. Η ομάδα του ΟΑΘ 29 χαιρετίζει την διαφάνεια των διαδικασιών των Αμερικανών. Έχει εκφράσει ωστόσο και ορισμένε επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των σχετικών δεσμεύσεων αλλά και την ασυμβατότητα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την συμβατότητα του ασφαλούς λιμένα. Πρώτα, για την έλλειψη απαρτίας στο Pay Club που είναι αυτή η οποία εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις που δεν επιτρέπει τους εποπτικούς οργανισμούς να εκτελούν το έργο τους. Η έκθεση επίσης και η συμπερίληψη στην έκθεση αυτή σχετικά με τους στόχους, με αυτούς που επιλέγουν, στο πρόγραμμα Upstream, αλλά και για τον, ε, την εκτελεστική διαταγή 1233. Επίσης, με συγχωρείτε μια στιγμή να διαβάσω καλύτερα, αυτό που είπε η ομάδα του άρθρου 29 στη γνωμοδότησή της του Ιουλίου 2016 είπαμε, είπαμε ότι δεν έχουμε επαρκείς αποδείξεις και νομικά δεσμευτικές που ε, να βεβαιώνουν ότι η συλλογή και η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από βάση Αμερικανικών αρχών δεν ε, σημαίνει μια ε, άνευ διακρίσεων πρόσβαση. Το ίδιο για τις προσφυγές των ενδιαφερομένων, που είναι σημαντικό κριτήριο που θεσπίζει στην απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για να υπάρχει επαρκής προστασία. Εμείς υπενθυμίζουμε ότι το κριτήριο standing requirement προσβασιμότητας της Αμερικανικής ε, νομοθεσίας προβλέπει μια δύσκολο να εφαρμοστεί προσφυγή από τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι προσφυγές που προσφέρονται στους ε, Ευρωπαίους πολίτες είναι περίπλοκες και δύσκολες και ο συνήγορος του πολίτη παίζει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την πρόσβαση για ζητήματα εθνικής ασφαλείας και προβλέπει το Privacy Shield, ακόμα δεν έχει οριστεί από τις Αμερικανικές Αρχές. Στην στη βάση αυτής της πρώτης ετήσης αξιολόγησης, το G29 ζητεί από τις Αμερικανικές και τις Ευρωπαϊκές Αρχές να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους και χωρίς καθυστέρηση να προχωρήσουν στη θέσπιση ενός σχεδίου δράσεως για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Αυτό το σχέδιο δράσεων θα βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ξεκάθαρο, που θα απαιτεί από τις Αμερικανικές αρχές να προβλέπουν τα δέοντα. Μέχρι τις 25 Μαΐου 2018 και την ε, θέση σε ισχύ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού απαιτούμε τον ορισμό συνηγόρου, ombudsman, ombudsperson αν θέλετε καλύτερα, και μέχρι την επόμενη ετήσια αξιολόγηση, δηλαδή το αργότερο τέλη του 2018, οι ελλείψεις και αβεβαιότητες που έχει εντοπίσει το G29 θα πρέπει να έχουν αντιμετωπιστεί. Αυτό που λέει το G29 επίσης είναι ότι εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση στην έκφραση των ανησυχιών και στις δύο προθεσμίες που έχουμε ζητήσει, οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα και ενδεχομένως και με προσφυγή στην εθνική δικαιοσύνη, που μπορεί πλέον από τον ε, Μάιο του 2018 να γίνει. Η έκθεση λοιπόν αυτή έχει ε, δημοσιευτεί και τώρα πού βρισκόμαστε αυτούς τους λίγους μήνες μετά από την έκφραση αυτών των επιφυλάξεων. Υπάρχουν και κάποια θετικά μηνύματα, αλλά και κάποια μάλλον αρνητικά. Σε ό,τι αφορά τα θετικά μηνύματα, βλέπουμε κάποια κίνηση από πλευράς Αμερικανικών αρχών γύρω από το θέμα της ε, έγκρισης του P-Club και του FTC. Εκτός όμως από αυτή τη δραστηριοποίηση και από τα πρόσωπα που ενδεχομένως να κατέλθουν υποψήφια, δεν έχουμε συγκεκριμένο διορισμό. Σε ό,τι αφορά τα μάλλον αρνητικά ε, μηνύματα, πρόκειται για την επανέγκριση από το Αμερικανικό Κογκρέσο του 700 2 του ΦΙΖΑ για άλλη μια εξαετία. Αυτή η εκ νέου έγκριση χωρίς καμία σημαντική αλλαγή σε ό,τι αφορά την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μη Αμερικανών πολιτών δεν είναι καλό σημάδι. Πρόκειται για κυρίαρχη απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου που μπορεί να θεωρηθεί σαν μια χαμένη ευκαιρία. Διότι ο G29 στην έκθεσή του προβλέπει πολλές συστάσεις για την παρούσα ε, νομοθετική θητεία, για το πρόγραμμα του 700, ε, του άρθρου 700 του ΣΦΙΝΤΑ, γιατί λέμε αντί να επιτραπεί η λειτουργία αυτού του προγράμματος επαγρύπνησης θα πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη στόχευση καθώς και εφαρμογή κριτηρίων όπως ε, δικαιολογημένες υποψίες για μια συγκεκριμένη ομάδα, ώστε αυτή να γίνεται αντικείμενο παρακολούθησης από μια ανεξάρτητη αρχή. Έχουμε λοιπόν, θα είδατε κι εσείς, όπως σας είπα, κάποια θετικά μηνύματα, αλλά και κάποια μάλλον ανησυχητικά. Εν τέλει όμως, ε, ποιο είναι το διακύβευμα που θεωρούμε ότι υπάρχει πίσω από την ασπίδα προστασίας Privacy Shield. Πρώτον, να αποδειχθεί αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού μοντέλου για την προστασία και μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε ένα πλαίσιο όπου οι ροές προσωπικών δεδομένων γίνονται όλο και πιο παγκοσμιοποιημένες. Ταυτόχρονα όμως ένας καθορισμός διεθνούς παγκόσμιου προτύπου. Και αυτό το παγκόσμιο πρότυπο τις επόμενες ημέρες και μήνες θα λάβει πλέον επιχειρησιακή σημασία που είναι προφανής και μάλιστα μέσω της εμπορικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προσανατολίζεται σε ένα, σε ένα πολλαπλασιασμό νέων συμφωνιών βεβαίως σε αυτά θα πρέπει να προβλεφθούν τα σχετικά μέτρα και μιλώ για συμφωνίες με την Ιαπωνία και την Κορέα. Η επεξεργασία και το επίπεδο των ε, προτύπων καταλληλότητας είναι απόλυτα καθοριστικά και θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη διάσκεψη του G29 Στι αποφάσεις αυτές θα περιληφθούν όλα τα στοιχεία που κρίνουν εάν η προστασία που χορηγείται σε τρίτη χώρα είναι επίπεδου συγκρίσιμου με το επίπεδο προστασίας που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και βεβαίω θα τα κρίνουμε αυτά με ρεαλισμό και θα προσαρμόσουμε το έγγραφο στη βάση των πληροφοριών που θα λάβουμε με, από τις συζητήσεις γύρω από την ασπίδα προστασίας. Αντιλαμβάνεστε κύριε Πρόεδρε ότι για το πρώτο αυτό θέμα έχουμε, ε, όπως είπα, τις πληροφορίες αυτές. Δεύτερο, η εφαρμογή του RGPD που είναι σημαντικό για την προστασία των δεδομένων. Το G29 εδώ και δύο χρόνια έχει ε, αποβεί πολύ δραστήριο στην παρακολούθηση αυτού του σημαντικού στόχου. Έχουμε καθορίσει ένα στρατηγικό σχέδιο δράσεως για το 2016 και 2020 για την εφαρμογή σε μια επιχειρησιακή πραγματικότητα και για τα άτομα και για τις οργανώσεις και για τις αρχές προστασίας δεδομένων. Πάνω από 20 ολομέλειες διεξαγάγαμε δηλαδή γύρω από το θέμα αυτό του γάμα δέλτα και 165 συνεδριάσεις τεχνικών υποομάδων είτε για το ένα είτε για το άλλο θέμα. Άρα, προς Θεού, αντιληφθείτε ότι το G29 υπήρξε πάρα πολύ δραστήριο στην παρακολούθηση της εφαρμογής του ΓΚΠΔ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων με ναι, επίση έγκριση πολλών κατευθυντήριων γραμμών ε, για συγκεκριμένα θέματα του κειμένου όπως η δυνατότητα μεταφοράς, όπως ο εντεταλμένο στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, το, τη δημιουργία προφίλ, την συνένεση, μέτρα διαφάνειας καθώς και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Εργασία η οποία γίνεται σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και με τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών μέσα από δημόσιες διαβουλεύσεις τις οποίες έχουμε διεξαγάγει και ε, με τα λεγόμενα Fab Lab. Και προσεγγίζουμε έτσι περισσότερο α, τις ανάγκες των χρηστών του κειμένου. Η δράση μας και στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο στρέφεται τώρα στην παρακολούθηση σε όλες τις χώρες μέλη, στην συνόδευση δηλαδή των προσπαθειών αυτών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή των αρχών του κανονισμού. Επειδή είμαι και πρόεδρος του G29, έχω δεσμευτεί η ομάδα μας να εγκρίνει και να δημοσιεύσει όλες αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και μάλιστα πριν από τον Μάιο του 2018. Όμως δεν θα σας κρύψω σήμερα, επειδή εκπροσωπώ τις διαφορετικές ευαισθησίες ε, στο ε, ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι αντιμετωπίζουμε και κάποιους τόνους που δεν είναι πάντοτε θετικοί η ρητορική γύρω από κάποιο εμπόδιο ε, στην πρόοδο. Δηλαδή, αυτά τα επιχειρήματα που ακούγονται. Απαντούμε στα επιχειρήματα αυτά με διαφόρους τρόπους. Και πρώτον, λέμε καθαρά ότι χρειάζεται ε, κάποιοι ε, να, γίνει μια προσπάθεια να προλάβουμε κάποια πράγματα. Κάποιοι οποίοι υστερούν και οι οποίοι δεν σέβονται αναγκαία σήμερα τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η οδηγία 1995, 1995. Δεύτερον, για το ΚΚΠΔ. Απαντούμε ότι ο ΚΚΠΔ φέρει τους Ευρωπαίους σε, επίπεδο, σε ίσο επίπεδο ανταγωνισμού με τους ε, παγκόσμιους φορείς σε ό,τι αφορά την στόχευση. Οι επόμενοι μήνες θα στραφούν γύρω από την παρακολούθηση εφαρμογής του ΚΚΠΔ, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Απαντούμε δε ότι το νέο δίκαιο που προβλέπει ο ΚΚΠΔ και ιδίως το δικαίωμα της μεταφοράς θα επιτρέψουν σε νέους φορείς να αναφιούν, θα επιτρέψουν ένα ρεύμα καινοτομίας και παροχής προσφοράς νέων υπηρεσιών και από νέους φορείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι όταν μιλούμε για το δικαίωμα μεταφοράς, καμία πλατφόρμα, ούτε αμερικανική, ούτε αλλοδαπή, δεν μπορεί να κρατά πλέον τον χρήστη και τα δεδομένα του. Μέσα από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στοιχηματίσει στην προστασία της προσωπικής ζωής ως ατού ανταγωνισμού. Αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε το στοίχημα αυτό και να γίνει και τρόπο ζωή. Άλλο σημαντικό που ήθελε ο νομοθέτης ήταν η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών. Ο Ευρωπαϊκό Κανονισμό προβλέπει ένα νέο μοντέλο διακυβέρνηση, το οποίο επιβάλλει στις, ε, ενδυναμώνει μάλλον τις ε, ευρωπαϊκές εθνικές αρχές, αλλά και τους επιτρέπει τη συνεργασία. Ο δε ε, μελλοντικός COPD που θα διαδεχτεί το G29 θα επιτρέψει περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην εφαρμογή του κανονισμού και πιο συγκεκριμένα δίνουμε τελική μορφή πλέον στους διαδικαστικούς κανόνες του ΚΚΠΔ και στους τρόπους και διαδικασίες της διαδικασίας του άρθρου 65 για την ρύθμιση διαφορών από την Επιτροπή. Και έχουμε και πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ ΚΚΠΔ και του Ευρωπαίου ε, εντεταλμένου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσει ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας που προβλέπει ο κανονισμός. Αυτή η νέα διακυβέρνηση είναι στοιχείο κλειδί για την επιτυχία του ΚΚΠΔ. Πρόκειται για την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του ρυθμιστικού μας μοντέλου, του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού μοντέλου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν δεν λειτουργήσει ο καινούριο COPD, όποια και να είναι, όποιες και να είναι οι αρετές του νομοθετικού κειμένου δεν θα επαρκέσουν. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι η συγκεκριμενοποίηση του νέου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων συνεπάγεται ότι οι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζουν ότι οι εποπτικές αρχές διαθέτουν τα αναγκαία μέσα κάθετος πόρους για να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα σε πολλές χώρες Η κατάσταση ωστόσο είναι πολύ διαφορετική. Μας φαίνεται λοιπόν σκόπιμο να μεταφέρουμε τον προβληματισμό αυτό ενώπιον των, των οφθαλμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ζητήσουμε να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Ορίστε κύριε Πρόεδρε, αυτά πολύ σύντομα είναι τα στοιχεία που μπορώ να θέσω υπόψη σας και για το G29 και για τον ΓΚΠΔ. Ευχαριστούμε πολύ Ιζαμπέλ. Ο λόγος τώρα στα μέλη. Κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μόλις προηγουμένως σήμερα το απόγευμα συζητούσαμε τη συνάδελφο Σιλβίγκη και έχουμε κάποιες ε, κοινέ ιδέες που θα ήθελα να σας ρωτήσω από πλευράς μας. Λέτε για επικριτικά σχόλια από κάποια από τα κράτη-μέλη. Όμως, γενικώς, πρέπει να πω ότι κάπως ενοχλούμε επειδή έχουμε μια νομοθετική πράξη που έχουν συναποφασίσει κοινοβούλιο και συμβούλιο και μπορεί να μην μας αρέσει, δικαίωμα του καθενός είναι, αλλά από τη στιγμή που έχει εγκριθεί και αποφασιστεί, καλό είναι να υλοποιείται. Ανησυχώ λιγάκι που τα κράτη-μέλη φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη από αυτού. Και με αυτή την παρατήρηση και έχοντα το κατά νου, ανησυχούμε επίσης που βλέπουμε ότι μόνο δύο κρατημέλη έχουν προσαρμόσει την εθνική τους νομοθεσία στον ε, γάμα κάπα Τι σημαίνει αυτό για την εφαρμογή που θα πρέπει να γίνει ως τον Μάιο του 2025 Μαΐου φέτος. Επίσης μια επιπλέον ερώτηση Είναι αλήθεια ότι όλα τα κρατημέλη έστειλαν τις απαραίτητες πληροφορίες στους πολίτες και τους ενδιαφερομένους ή μόνο τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και να κάνουν τους σχετικούς ελέγχους αν θέλουν να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Και τελευταία ερώτηση. Τι μπορούν να κάνουν οι περιφερειακές αρχές των κρατών μελών για να υποστηρίξουν τους αρμόδιους και να δώσουν και περισσότερες πληροφορίες στους πολίτες. Προσωπικά θα ήθελα μια δική μου ερώτηση να θέσω για την ασπίδα προστασία της ιδιωτικότητας. Είπατε ότι υπάρχει κάποια πρόοδο σε σχέση με την ε, προηγούμενη φάση και ότι είναι μια βελτίωση σε σχέση με τον ασφαλή λιμένα όταν όμως κοιτάζω τι πρόοδος έχει επιτελεστεί ως προς την υλοποίηση της ασπίδας προστασίας, έχω κάπως την εντύπωση ότι είναι μια επανάληψη της διαδικασίας του ασφαλούς λιμένα. Διότι ούτε όλα υλοποιούνται και οι Ηνωμένε Πολιτείες κάνουν πολύ βραδία πρόοδο. Αναφέρατε το τι λείπει από το P-Club, το ίδιο γινόταν και με το FISA, παρευλήματα που μας έχουν μείνει από το παρελθόν. Άρα το ερώτημα είναι όσο ομάδα εργασία του άρθρου 29 εσείς τι μπορείτε να κάνετε για να παραμείνει αμύωτη η πίεση και να υλοποιηθούν κάποια πράγματα. Πιστεύετε ότι και εμείς ως κοινοβούλιο μπορούμε να απαιτήσουμε ε, ότι ό,τι έχει εγκριθεί ως απόφαση να υλοποιηθεί στο συντομότερα. Ευχαριστούμε, Μπίργκιτ, η κυρία Ιντβελτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Φάλκε, Πιερωτά, για την ε, εισήγησή σας. Πολύ σύντομα για τον γάμα κάπα πι Συμφωνώ με την προηγούμενη ομιλήτρια. Δεν μπορούμε να δεχτούμε καθυστερήσεις και στα Ολλανδικά μέσα Άκουσα ότι οι ενώσεις ζητούν αναβολή. Εάν ξεκινήσαμε τη δουλειά για αυτή τη δέσμη το 2011, ε, εάν ζούσαμε στην εποχή του λίθου, δεν θα το ξέραμε ότι κάτι πήκεται. Το εγκρίναμε πριν δύο χρόνια. Είναι πολύ άδικο για αυτές τις εταιρείες και αυτούς τους οργανισμούς που έχουν ετοιμαστεί, έχουν κάνει τα μαθήματά τους και το έχουν υλοποιήσει, να μην απαιτηθεί άμεση δράση. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε αναβολέ να ανασκουμποθούν και να προλάβουν και οι υπόλοιποι. Για την ασπίδα προστασία δεν χρειάζεται να πω ότι πιστεύω ότι η ασπίδα αυτή δεν είναι νομικός αεροστεγής και ασφαλής και αν δείτε την υλοποίηση να πω ότι τον 1,5 χρόνο μετά τη θέση σε ισχύ ε, ένας μόνιμος ε, διαμεσολαβητής ακόμη δεν έχει οριστεί το P-Club δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύριος Άνταμ Κλάιν ε, ε, ορίστηκε από τον κύριο Τραμπ να αναλάβει το P-Club. Δύο από τους πέντε έχουν διοριστεί. Όμως το θέμα είναι ότι αν δούμε το ιστορικό του κύριου Κλάιν, το βιογραφικό του, έχει αντιταχθεί σε όλες τις μεταρρυθμίσεις του NSA. Τι είδους εμπιστοσύνη πρέπει μπορούμε να του έχουμε. Και τέλος, και αυτό είναι και το σοβαρότερό μου ερώτημα, η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή της ότι η επικείμενη συζήτηση για τα άρθρα 7,2 του ε, νόμου περί παρακολούθησης ενισχύουν το Κογκρέσο και το, ε, τη Βουλή σε όσα μπορεί να αποφασίσει σε σχέση με το ΦΙΖΑ και τα εργαλεία που αυτό προσέφερε βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι εγγυημένη η αναθεώρηση του άρθρου 702. Επίσης, ψηφίστηκε αυτό και η παράτασή του χωρίς καμία τροποποίηση τελικά. Και ε, πολύ ενδιαφέρον επίσης ότι μια μισή ώρα πέντε την ψηφοφορία έλαβα επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγοντας το Αμερικανικό Κογκρέσο μπορεί και να ψηφίσει για το θέμα αυτό. Τι είδου παιχνίδι είναι αυτό. Δεν λέω να απαντήσετε εσεί οι ίδια, αλλά έπρεπε να το πω εδώ. Διότι ειλικρινώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει παιχνίδια τέτοιου είδου. Είναι λίγο προσβλητικό να λαμβάνει κανεί τέτοια επιστολή ε, μια μισή ώρα πριν την ψηφοφορία. Είναι προσβλητικό προ αυτό το σώμα και του πολίτε τη Ευρώπη. Πώ να σα εμπιστευόμαστε έστω και λίγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, που υποτίθεται ότι παρακολουθείτε ως θεματοφύλακες την υλοποίηση του, της ασπίδας προστασίας, τουλάχιστον μέχρι να την ε, κηρύξουν άκυρη τα δικαστήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που βλέπω να υπάρχει και ανάλυση και ο δικός χάρτης για το πώς θα προχωρήσουμε. Είναι σημαντικό με νέους νόμους ε, τα πρότυπα του ΓΚ δέλτα, πι δέλτα να ισχύουν, διότι εάν μετά τις 25 Μαΐου οι βελτιώσεις δεν έχουν ενσωματωθεί, δεν έχουν επιτευχθεί, θα πάμε στα δικαστήρια. Συμμερίζομαι τις μέρημνες των συναδέλφων και δεν θέλω να επαναλάβω όλα όσα είπαν ως ανησυχίες τους. Απλώς να θέσω κι εγώ μια επιπλέον ερώτηση που αναφέρεται στην υπόθεση της Microsoft ε, όπου δικάστηκε στο το Δικαστήριο και το ερώτημα εν τέλει είχε να κάνει με την πρόσβαση της αστυνομίας στα δεδομένα. και αν αυτό έχει κάποια επίδραση στην ε, πράξη, την απόφαση περί ε, και αν το άρθρο 29 το συζήτησε αυτό. Εσείς ως ομάδα του άρθρου 29. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να ασκήσουμε περισσότερη πίεση για να βελτιωθούν τα πρότυπα του, της ασπίδας προστασίας. Η ερώτηση νομίζω συχνά ανακαιτεί και εύλογα για το κατά πόσο είμαστε το ίδιο αυστηροί με τα κράτη-μέλη και τη δική τους προστασία. Υπάρχει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Δεκεμβρίου 2016 που δεν έχει εφαρμοστεί στα 28 κράτη-μέλη. Για να είμαστε λοιπόν πιστικοί ως προς την υλοποίηση μέχρι τις 25 Μαΐου. Καλό θα ήταν οι υπεύθυνοι να φροντίζουν και για την εφαρμογή της νομολογίας του ΔΕΚ όταν ε, μιλάμε για τα κρατη και τα μέτρα παρακολούθησης κατά μελών που δεν συμβαδίζουν και δεν ακολουθούν τις αποφάσεις του ΔΕΚ. Ευχαριστούμε Γιάννη. Αναγκόμες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Να υπογραμμίσω το ότι έχει σημασία ο διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι ανεξάρτητος. Δεν ισχύει αυτό στο παρελθόν. Είναι ένα θέμα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιμείνει. Μετά από τις αποφάσεις της πρόσφατες της FCC, για την κατάργηση της ουδετερότητας του δικτύου, το net neutrality. Αυτό δίνει πλήρη έλεγχο στις μεγάλες επιχειρήσεις και είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα στην φορητότητα. Και τέλος, Αναφερθήκατε στην ρητορική, την ενοχλητική και για σας από ό,τι κατάλαβα. Για το πλαίσιο, το δεσμευτικό, η οποία υπάρχει όχι στις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιος άλλος θα ήθελε το λόγο. Ζητώ πρώτα συγγνώμη διότι δυστυχώς καθυστέρησα να φτάσω και δεν άκουσα την παρέμβαση της εκπροσώπου. Η κατάσταση ωστόσο είναι σχετικά σαφής. Με συγχωρείτε λέει ο κ. Βόσνε, ναι, σας διέκοψα γιατί συνομιλούσατε με τον διπλανό σας. Είναι σαφής η κατάσταση, επαναλαμβάνω. Έχουμε την ε, ασπίδα προστασίας που υποτίθεται ότι είναι βελτίωση του ασφαλούς λιμένα και επίσης εφαρμόζει τα κριτήρια της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και επίσης έχει υποτίθεται τον χαρακτήρα να επιτρέψει ένα γενικότερο έλεγχο και εκτός από αυτό να βελτιώνεται διαρκώς ο έλεγχος. Αυτό πάντοτε θεώρησα εγώ ότι ε, είναι το σωστό. Δηλαδή ξεκινεί κανείς με το Privacy Shield και μετά βλέπει πώς αυτό μπορεί να συμπληρώνεται σταδιακά. Τώρα έχουμε απέναντί μας μια Αμερικανική διοίκηση η οποία δεν ανταποκρίνεται ας πούμε ακριβώς σε αυτά που θεωρήσαμε ότι θα ισχύουν τότε όταν τα κάναμε όλα αυτά. Το ερώτημα είναι εάν πράγματι πρόκειται για έλλειμμα ή εάν εν πάση περιπτώσει τα όσα διαμορφώνονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού όντως θα οδηγήσουν στην πρόοδο που αναμένουμε. Το ερώτημα που έχω εγώ είναι κατά πόσον αυτό μπορεί όντως να προκαλέσει νομικά μειονεκτήματα για το μεμονωμένο άτομο. Χρειάζεται μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση, αλλά από γενική σκοπιά θα πρέπει να είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε ένα θεμέλιο για την ανταλλαγή ε, αυτή δεδομένων. Έχουμε καθορίσει κάποια κριτήρια, τα οποία υποτίθεται ότι θα βελτιώνονται διαρκώς και ότι εάν υπάρχει ένα έλλειμμα, και το έλλειμμα είναι δύσκολο να καλυφθεί εφόσον δεν προχωρά η Αμερικανική διοίκηση, το ερώτημα είναι κατά πόσον αυτό αποτελεί μειονέκτημα. Καταρχήν δεν μας αρέσει βέβαια αυτό που κάνει η Αμερικανική πλευρά, αλλά ποια είναι τα μειονεκτήματα εν τέλει. Εξάλλου, το ερώτημα πάλι είναι ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν παραπέρα ή ποια μέτρα που μπορούν να ληφθούν μπορούν να δημιουργήσουν σε βελτίωση γύρω από αυτό στρέφεται η δική μου σκέψη. Διότι να ανακοπεί ή και να διακοπεί η μεταφορά δεδομένων, ε, νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα. Χρειάζεται βελτίωση. Γι' αυτό θα ήθελα να μάθω τι μπορεί να γίνει ως συγκεκριμένη βελτίωση. Θέλετε να επανέλθετε, κύριε Σίπελ. Ναι, ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε όχι τόσο ως ερώτηση, αλλά πιο πολύ μια σύντομη παρατήρηση. Εάν προχωρούμε σε σύναψη διεθνούς συμφωνίας, θεωρώ ότι όλα τα μέρη, όλα τα συμβαλόμενα μέρη έχουν την ίδια σημασία και δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στους εταίρους μας να πούμε «Α, αυτό το τμήμα της εννοεί τμήματα τη Αυτό το τμήμα της συμφωνία είναι σημαντικό, θα το εφαρμόσω. Άλλο τμήμα της συμφωνίας δεν είναι σημαντικό, δεν θα το εφαρμόσω. Όχι, όλα τα τμήματα της συμφωνίας θα πρέπει να εφαρμόζονται και αυτά θα πρέπει να αποτελούν την βάση για την διαρκή επανεξέταση και για να απαιτηθεί απέναντι στις Αμερικανικές Αρχές να τηρούν απολύτως τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Ναι, θέλω και εγώ μια ερώτηση να κάνω για το γενικό κανονισμό. Και τι θα κάνουν τα εθνικά κοινοβούλια στο Μάιο. Ε, μπορεί να γίνει δίκοπο μαχαίρι όσο και αν είναι σημαντικό να προλάβουμε την υλοποίηση. Εάν δεν έχουν γίνει οι κινήσεις που πρέπει και δεν είναι πλήρης οι προσαρμογές. Μπορείτε λιγάκι να μας το προσδιορίσετε. Όχι αναγκαστικά προς την εφαρμογή της νομοθεσίας. Εκεί που εφαρμόζεται ήδη η νομοθεσία, ας πούμε, και υπάρχουν άλλοι φραγμοί. κάποια αντίσταση από τις εταιρείε, διότι καταλαβαίνουν ότι αυτό που μπορεί να συμβεί είναι οι καταναλωτές να παίρνουν περισσότερες πληροφορίε. Μας λέτε πώς το βλέπει η Επιτροπή του Άρθρου 29. Τι σημαίνει στην παρακολούθηση και την εξέλιξη της ε, υλοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για την ασπίδα προστασίας. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι η ασπίδα προστασίας είναι πρόοδο σήμερα σε σχέση με τον ασφαλή λιμένα. Οι Αμερικανοί την έλαβαν σοβαρά υπόψη την υπόθεση και υιοθέτησαν πλήρη, πλήρη σύστημα για την πλήρη υλοποίηση του Privacy Shield, τη στιγμή, πράγμα που δεν υπήρχε τη στιγμή υιοθέτηση του Safe Harbor. Υπάρχει λοιπόν σαφής πρόοδος με την ασπίδα σε σχέση με το λιμένα. Πέραν αυτού λείπουν κάποια στοιχεία για τα οποία εκφράσαμε επιφυλάξεις. Η θέση που τήρησε η ομάδα του άρθρου 29 είναι ρεαλιστική από το μήνα Οκτώβριο κιόλα. Δηλαδή, να συμπαρασύρουμε τους Αμερικανούς σε μία πορεία προόδου, ορίζοντάς τους ένα χρονοδιάγραμμα σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα είναι τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν σχετικά εύκολα και γρήγορα, μέτρα επάνδρωσης, το P-Club, ο διαμεσολαβητής, ο ή η διαμεσολαβητής, διαμεσολαβήτρια. Εδώ δεν υπάρχουν βασικά νομικά προβλήματα, είναι θέμα απόφασης που πρέπει να ληφθεί. Και μας φάνηκε ότι συνδυάζοντας αυτό το πρόγραμμα δράσης που ζητούμε από τις Αμερικανικές Αρχές, ε, βρισκόμαστε σε μια λογική πραγματιστική, διότι αυτό που ζητάμε για τον μήνα Μάιο δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει και γιατί κατά τα άλλα συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση που είχαμε ασκήσει και τη στιγμή του ασφαλούς λιμένα, ώστε το σύνολο του συστήματος να προχωρεί ως προς τους διορισμούς. Καταλαβαίνουμε ότι το αίτημα προς τις Αμερικανικές αρχές ε, έγινε, εισακούστηκε, διότι ως προς τους διορισμούς ε, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Εγώ έχω βάσιμες ελπίδες ότι ως τον Μάιο θα έχουμε ανθρώπους που θα προσληφθούν όντως για αυτές τις θέσεις. Τώρα, αν επί της ουσίας αυτό θα είναι αρκετό, κατά πάσα πιθανότητα όχι. Και όταν με ρωτάτε, μεν και δε, τι μπορούμε να κάνουμε για να παραμείνει η πίεση, νομίζω το Κοινοβούλιο πρέπει να ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση και να επιμείνει στα θέματα ουσίας, ε, όπως είχε κάνει αρχικά η ομάδα του άρθρου 29. Αυτό είναι πλέον έκτημα ή μειονέκτημα για τους Ευρωπαίους. Να σας πω Αυτό που χρειάζονται οι Ευρωπαίοι αλλά και όσοι φορεί ασχολούνται με αυτά τα δεδομένα χρειάζονται ένα νομικό πλαίσιο που να είναι εύρωστο, το οποίο να μην είναι θύμα οποιασδήποτε δικαστική προσφυγή και θα οδηγούσε σε ακύρωση, αναστολή του συστήματο. Αυτή τη στιγμή ισχύει αυτό. Έχουμε δύο προσφυγέ τουλάχιστον στα δικαστήρια να εκδικάζονται και ειλικρινώ δεν ξέρουμε ποια θα είναι η έκβασή του. Δεν ξέρουμε τι απόφαση αυτό που λέμε εμείς λοιπόν στο επίπεδο της ομάδας του άρθρου 29 είναι ότι αυτή τη στιγμή ε, αρνούμαστε εμπορικέ ε, διαπραγματεύσεις με μεγάλες χώρες και χρειαζόμαστε ε, μια απόφαση προσαρμογής που να είναι πραγματικά εύρωστη με ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον για αυτό το πρότυπο, ας εκμεταλλευτούμε τα διδάγματα που αντιλήσαμε από τις διαπραγματεύσεις για την ασπίδα και ας δούμε τι επίπεδο θέλουμε να έχουμε τουλάχιστον στην Ευρώπη. Όλα αυτά αποτελούν ύλη που δεν είναι πυρηνική φυσική. Δεν είναι επιστημονικά όλα αυτά. Βλέπουμε ότι προχωρούμε βήμα-βήμα. Και βλέπουμε ότι βήμα-βήμα ακριβώς ε, οδηγούμε τους Αμερικανούς και τις τρίτες χώρες να προσφέρουν εγγύησει που εμείς οι Ευρωπαίοι τις ε, θέλουμε. Αλλά νομίζω ότι όσο παραμένουμε σε αυτή την δυναμική πορεία και την πρόοδο προ το μέρο μα αυτών των τρίτων χωρών, το θεωρώ θετικό. Για την ώρα πάντω η στρατηγική αυτή έχει δώσει αποτέλεσμα στο επίπεδο τη ομάδα του άρθρου 29 και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Τώρα για το Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων. Για το Γενικό Κανονισμό. Η μουσική κριτική που ακούγεται σε σχέση με τα κράτη-μέλη και εκφράζει τη δηλία κάποιων κρατών μελών, η δηλία αυτή σε σχέση με το νομικό πλαίσιο είναι κάτι που εμάς μας περιορίζει. Βεβαίως δεν είναι σωστό, αλλά πρέπει να ακούσουμε μεν τι έχουν να πούν ε, Πρέπει να ακούσουμε τα διάφορα επιχειρήματα και να απαντήσουμε. Ε, για τα κράτη. Εάν τα κράτη είναι σε κατάσταση να προχωρήσουν και να συγκλίνουν ως προς το γενικό κανονισμό. Όχι. Δεν είναι αμέσως, διότι το, ο γενικός κανονισμός προβλέπει τουλάχιστον 50 ε, αλλαγές σε εθνικές νομοθεσίες αλλά είναι επιλογή. Δεν χρειάζεται να γίνει μέσω εθνικής νομοθεσίας η εφαρμογή του ΓΚ. Ε, είναι κανονισμός, όχι οδηγία, εκτός από μία περίπτωση. Αυτά που έχουν να κάνουν με τις εθνικές αρχές των εθνικών κρατών. Αυτό που είναι τελείως καινούργιο σε σχέση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων είναι η διαδικασία συναπόφαση που προβλέπει τη συνάρθρωση των ε, ε, εθνικών κατασταλτικών αρχών, δράσεων μάλλον, με τις δράσεις διαμεσολάβησης της νέας επιτροπής που θα αντικαταστήσει την ομάδα του άρθρου 29. Αν όμω οι εθνικοί νομοθέτε δεν το επιθυμήσουν αυτό, αυτό το συνδυασμό, αυτή τη συνάρθρωση, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται αυτή η εθνική παρέμβαση για να τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμό. Σε επίπεδο όμω ομάδα άρθρου 29, ε, δείξαμε την απαραίτητη προσοχή για να είμαστε βέβαιοι ότι η εναρμόνιση που απαιτεί ο κανονισμό γίνεται εντό τη περίοδου που ακολουθεί. Γι' αυτό και στις κατευθυντήριες γραμμές εντοπίσαμε τα σημεία κλειδιά, τις έννοιες κλειδιά του νέου ΓΚΠΔ, ώστε οι αρχές προστασίας των δεδομένων να συμφωνήσουν για κοινέ θέσεις, ώστε να αποφύγουμε η μεν ή η δε να ε, Δηλήσουν ε, με την εθνική μετάφραση σε νομοθεσία τον γενικό στόχο του κανονισμού. Αυτά ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές. Τερναίο, τε, τελευταίο, τελευταίο στοιχείο για τον ε, γάμα πιδέλτα και τις εθνικές αρχές. Πώς μπορεί να γίνει ένα ατού της Ευρώπης αυτός ο κανονισμός και όχι πατερίτσα. Ε, εγώ συμφωνώ ότι πρόκειται για τούτη τη Ευρώπη φυσικά και ότι από την άποψη του νομικού πλαισίου μπορεί να μα βοηθήσει να χρησιμοποιήσουμε τι νομικέ προσφυγέ ω ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μέσω των στρατηγικών παρακολούθηση και τα εργαλεία που οι αρχέ εφαρμογή θα θέσουν στη διάθεση των ε, φορέων στου διάφορε χώρε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα το πετύχουμε αυτό. Σε μερικέ χώρε, τα εργαλεία αυτά υπάρχουν ήδη για τι μικρομεσαίε επιχειρήσεις και τα εργαλεία αυτά τα έχουμε φέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε και πάλι να έχουμε μια στρατηγική παρακολούθησης που να είναι εναρμονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεδομένων των στοιχείων αυτών, πιστεύω ότι ο στόχος των ερχών προστασίας δεδομένων μπορεί να ακολουθήσει αυτών των Ευρωπαίων φορέων στα πλαίσια του νομικού πλαισίου. Ω προ τη στρατηγική, την κατασταλτική στρατηγική, τη στρατηγική καταστολής, είναι μεγάλο ο αριθμό των υπευθύνων που έρχονται να μα δουν και μα λένε τι θα γίνει το Μάιο τελικά. Θα επιβάλλεται κυρώσει σε όλου. Όσοι δεν συμμορφώνονται με το γενικό κανονισμό θα τιμωρηθούν. Όσοι έχουν καθυστερήσει με τι νέε υποχρεώσει. Εγώ το έχω πει επανειλημμένω και το ξαναλέω και μπροστά σα. Για μα δεν είναι λεμιτόμο το γενικό κανονισμό. Δεν θα επιτεθούμε σε όλου του υπευθύνου ε, το Μάιο και να του τιμωρήσουμε για τι υποχρεώσει που δεν έγιναν σεβαστέ. Θα ακολουθήσουμε μια στάση μαθησιακής καμπύλης και μαθησιακών καμπυλών εφόσον ε, απαιτηθεί αυτό Ε, πάντως για τις αρχές του γενικού κανονισμού, τα εργαλεία είναι καινούργια αλλά όχι αρχές. Είναι οι ίδιες αρχές που υπήρχαν και στην οδηγία του 95. Οι αρχές του τελικού σκοπού της αναλογικότητας, εντάξει τα ελέγχουμε και τα παρακολουθούμε, από τον Μάιο θα αρχίσει ο έλεγχος, αλλά ήδη κάνουμε αυτόν τον έλεγχο σήμερα. Ευχαριστούμε Ιζαμπέλα, αλλά σοφή γρήγορα παρακαλώ. Ναι, μια πρωτασούλα μόνο. Επειδή λέτε ότι δεν θα είμαστε παράλογοι στην επιβολή από τις 25 Μαΐου. Ναι, αλλά θέλω να ρωτήσω. Θα λάβουν υπόψη υπεύθυνοι του Γενικού Κανονισμού ότι κάποιοι οργανώ... κάποιες οργανώσεις και ενώσεις κατέβαλαν μια επιπλέον προσπάθεια, ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η διακεκριμένη διαφοροποίηση. Για όσους προσπάθησαν και τα έδωσαν όλα για να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Ενώ στη χώρα μου κάτι υπουργεία ακούω ότι δεν επένδυσαν καν το χρόνο και τα μέσα που έπρεπε. Δεν πρέπει κάτι να γίνει. Νομίζω ότι απάντησα ήδη. Οι ρυθμιστές νομίζω ότι είναι λογική ε, στην εφαρμογή. Ο στόχος δεν είναι να υπάρξουν τιμωρίες. Ο στόχος είναι όλες οι ευρωπαϊκές αρχές να ε, λάβουν τα μέτρα τους. Η τιμωρία είναι αποτρεπτικό μέτρο. Η Επιτροπή μας επιβάλλει 15 κυρώσεις ετησίως από 8.000 προσφυγές. Είναι πολύ εξαιρετικό εργαλείο αποτροπής. Δεν είναι μέσο για να ρυθμίσουμε την κανονικότητα και την καθημερινότητα. Αυτά θα είναι τα εργαλεία συμμόρφωσης και συμβατότητας που ήδη έχουμε προτείνει στους διάφορους φορείς και προφανώς θα λάβουμε υπόψη τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί ή όχι. Απλώς ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο εξής Μπορεί να είμαστε πάρα πολύ ευέλικτοι με τα εργαλεία, με το ότι είναι καινούργιο στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σε σχέση με την οδηγία του 1995 αλλά εάν πρόκειται για μια γενική αρχή που ισχύει από 20 ετία, εκεί θα θέσουμε διαφορετικά το ερώτημα. Thank you, Isabel. Thank you, um, for... Uh, Ευχαριστούμε, Ιζαμπέλ. Σας ευχαριστώ για την συνεισφορά σας σήμερα. Ότι στις 29 Φεβρουαρίου θα προεδρεύσουμε της ομάδας εργασίας. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Φάλ Πιερωτά για την εξαιρετική προσπάθεια την οποία έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί στενά, σας ευχαριστώ και ε, οι καλύτερες ευχές στην ομάδα σας. Νομίζω ότι πράγματι αυτά τα οποία μας είπατε σήμερα θα μας δώσουν την δυνατότητα να συζητήσουμε στην επόμενη συνάντηση το θέμα για την ασπίδα ασφαλείας και για το αν θα κάνουμε μια ε, έκθεση γύρω από αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την συνεισφορά σας. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την εξαιρετική συζήτηση. Οι ψηφοφορίες θα ξεκινήσουν σε, 11 λεπτά ακριβώς, σε 4 λεπτά ακριβώς. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Colleagues, uh, take your seats. We're going to go straight to the vote. Everyone take your seats. Καθίστε παρακαλώ αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Θα διεξαχθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία, γι' αυτό παρακαλώ πάρτε τις ηλεκτρονικές κάρτες και βάλτε, τις στην ε, ε, ενδεδειγμένη σχισμή. Αν δεν έχετε την κάρτα σας, παρακαλώ να μου το γνωρίσετε τώρα και θα σας σημειώσουμε για την ψηφοφορία. Ποιος δεν έχει ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορία. Υπάρχει κανείς που δεν έχει. Υπάρχει κάποιος εκ των βουλευτών που δεν έχει. Άρα τις έχετε όλοι. Καθίστε όλοι παρακαλώ και βάλτε τις κάρτες στην ε, σχισμή σας παρακαλώ πιο σύντομα. τη διάρκεια της συναντήσεως της 11ης Ιανουαρίου 2018 οι συντονιστές σημείωσαν την απόφαση της 20ης Σεπτεμβρίου 2017 της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, κίνηση του άρθρου 7 της συνθήκης κατά της ε, δημοκρατίας της Πολωνίας. Και οι συντονιστές συζήτησαν τα περαιτέρω θεωρώντας ότι είναι αναγκαίο ψήφισμα το οποίο να εκφράζει την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θεώρησαν ότι ε, μπόρεσαν μάλλον να το εγκρίνουν με πλειοψηφία οι συντονιστές σύμφωνα με στη βάση μόνο γραπτής διαδικασίας. Για διαδικαστικό θέλετε τον λόγο κυρία μου. Πέστε μου το όνομά σας σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να το διαβάσω δυστυχώς στην πινακίδα. Λέγομαι Γκοσεύσκα. Κύριε Πρόεδρε, έχω ένα διαδικαστικό θέμα, διότι στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ιστοσελίδα δηλαδή, ναι, ναι, σας παρακαλώ, σε λιγότερο από δύο λεπτά λέει ο Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται να ψηφίσουμε ψήφισμα για την Πολωνία. Έως τώρα στην ιστοσελίδα Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν υπάρχει πολωνική ιστοσελίδα, μόνο αγγλική και ο κανονισμός λέει ότι θα πρέπει να μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες εργασίας. Από πότε τα πολωνικά έπαυσαν να είναι επίσημη γλώσσα εργασίας τη Ένωση. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Πόσα διαδικαστικά θα μου υποβάλλετε σήμερα. Δύο. Άλλος κανεί, Εσείς κύριε Γιούρεκ, το δεύτερο διαδικαστικό. Και μετά θα απαντήσω και στα δύο. Σε σχέση με πληροφορίες που έλαβα στις 3 το απόγευμα, θα ήθελα να μου δώσετε κάποια δικαιολόγηση για το εν λόγω ψήφισμα, διότι και αν ακόμη υποστηριχθεί από κάποιους, δεν ξέρω από ποιους, αλλά ο πρόεδρος είπε ότι το υποστηρίζουν όλες οι πολιτικές ομάδες, σίγουρα δεν το υποστηρίζει η ομάδα των μεταρρυθμιστών ε, και συντηρητικών, αν και αν ακόμα υποστηριχθεί, οι συντονιστές θα πρέπει να προβάλλουν κάποιους λόγους για το ψήφισμα αυτό. Επαναλαμβάνω ότι η πρόταση που υπέβαλε η Κομισιόν στο Συμβούλιο περιλαμβάνει και την ανάγκη τοποθετήσεως με ενισχυμένη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα αυτή είναι η συνήθη διαδικασία για τέτοιο ψήφισμα. Ωστόσο εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο υποτίθεται ότι ψηφίζουμε σήμερα επί ψηφίσματος το οποίο δεν συζητήθηκε ποτέ. Ούτε καν η αιτιολόγησή του δεν ψηφίστηκε ποτέ. Θα ήθελα να ακούσω πρώτον την αιτιολόγηση και δεύτερον θα ήθελα να γνωρίζω εάν όντω το υποστηρίζουν όλοι οι συντονιστέ των πολιτικών ομάδων, διότι η δική μα ομάδα σίγουρα δεν το υποστηρίζει. Τέλο, εγώ θεωρώ ότι είναι περιττό, διότι με τον τρόπο αυτό διχάζεται η Ευρώπη. Με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι ατυχής, αλλά αυτή ακολουθήσει η διαδικασία. Ούτω ή άλλω, εγώ δεν τι κατανοώ τι διαδικασίε αυτέ. Γιατί πρέπει εμεί να, ψηφίσουμε και ε, ζητώ να αποσυρθεί ο πρόεδρο Κλοντ Μωρά. Και για την άλλη, απαντώ και στην άλλη ε, ευρωβουλευτή, τη οποία δυστυχώ δεν βλέπω το όνομα. Υπάρχουν άλλα διαδικαστικά. Αν υπάρχει άλλο διαδικαστικό, δεν θα μπορέσω να το ακούσω. Α, βλέπω ότι υπάρχει ένα διαδικαστικό ακόμη. Πρόκειται για διαδικαστικό κύριε. Ας τα ακούσουμε όλα. Ας τα ακούσουμε όλα. Πρώτα και μετά θα απαντήσουμε. Δύο λεπτά παρακαλώ. Μην υπερβείτε τα δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα την αιτιολογήση που δώσατε στις 3 το απόγευμα και προσπάθησα στο σημείο αυτό της ημερησίας διατάξεως υπαριθμών 5 να βρω το ψήφισμα. Πρόκειται για το 2541 του 2018 και όταν κανείς ψάχνει να το βρει αυτό στο διαδίκτυο βγαίνει στα αγγλικά μια φράση που λέει το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει το κείμενο αυτό, αν δεν το γνωρίζω, πώς θα ψηφίσω αφού ούτως ή άλλως καν δεν γίνεται συζήτηση γι' αυτό. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Άκουσα, νομίζω, με γενεοδορία ψυχής όλα τα διαδικαστικά σας. Ας αρχίσουμε τώρα από το τελευταίο. Όλα τα μέλη έχουν πρόσβαση στο κείμενο, το οποίο είναι δημοσιευμένο ήδη από τις 9 το πρωί. Τώρα, αυτά για τον κύριο Βόιτ πρώτον. Ο κύριος Γιούρεκ, είπα ορισμένα πράγματα προηγουμένως. Θα ξαναπώ τώρα, οι συντονιστές αποφάσισαν με πλειοψηφία για το ε, σχέδιο του κειμένου αυτού. Πρόκειται λοιπόν για απόφαση ληφθήσα κατά πλειοψηφία. Αυτό απαντά στην ερώτησή σας αν το υποστηρίζουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Γίνεται η ψηφοφορία και μετά θα ακολουθήσει πλήρη συζήτηση στην Ολομέλεια. Συζήτηση σήμερα δεν γίνεται, γι' αυτό γίνεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αυτή είναι η απόφαση των συντονιστών, επαναλαμβάνω, ελήφθη με πλειοψηφία. Η γλωσσική εκδοχή του σχεδίου είναι στα αγγλικά διότι αυτό δεν επιτρέπει περισσότερα το χρονοδιάγραμμα, θα υπάρξει βεβαίω πλήρης πολωνική μετάφραση για την Ολομέλεια. Ζητώ την άδειά σα για να προχωρήσω την ψηφοφορία. Δυστυχώς δεν μπορώ να δεχθώ άλλα διαδικαστικά. Πώς μπορούμε να ψηφίσουμε χωρίς να γνωρίζουμε το κείμενο. Θα απαντήσω άλλη μια φορά, απαντά ο κύριος Μωράης στην κυρία Κοσχεύσκα, λόγω του χρονοδιαγράμματος και επειδή είναι σχέδιο κειμένου, έχουμε την άδεια να προχωρήσουμε μόνο στη βάση του αγγλικού κειμένου. Θα υπάρξει πλήρης, πλήρης πολωνική μετάφραση για την Ολομέλεια. Θα προχωρήσω τώρα στην ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Άρχισε η ψηφοφορία. Has Ψηφίσατε όλοι και όλες. Η φιλελεύθερη ομάδα έχει μία πλεονάζουσα ψήφο. Παρακαλώ ρυθμίστε ώστε να αφαιρεθεί μία. Μάλιστα, έκλεισε τώρα η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 33 ψήφους ε, υπέρ, 9 κατά και καμία αποχή. Σας ευχαριστώ αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ έληξε η ώρα της ψηφοφορίας και θα γίνει η ψήφιση ε, στην Ολομέλεια του ε, Μαρτίου. Colleagues, the next part of the agenda is 1710. 1710. Um, Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο είναι σημαντικό και ενδιαφέρον, εάν μπορούν να παραμείνουν οι συνάδελφοι, εάν βεβαίως έχουν ε, έρθει μόνο για την ψηφοφορία και επιθυμούν να αποχωρήσουν, αλλιώς σας παραμείνουν, έχουμε την ακρόαση της υποψήφιας για την θέση του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπόλ. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε κοντά μας σήμερα την επιλεχθήσα υποψηφία Κατρίν Ντεμπόλ ε, η υποψηφία επιλεγμένη από το Συμβούλιο από κατάλογο υποψηφίων που έχει προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για την θέση εκτελεστικής διευθύντριας της Ευρωπόλ στις 23 Δεκάτου οι συντονιστές της ΛΥΜΠΕ αποφάσισαν να εφαρμόσουν το άρθρο 54 του κανονισμού 794-2016 για την Ευρωπόλ και να προσκαλέσουν την επιλεχθήσα υποψήφια για την θέση της αναπληρώτητας διευθύντριας της, ε, μάλλον, ε, συγγνώμη, της εκτελεστικής διευθύντριας της Ευρωπόλ, να προσκαλέσουν δηλαδή ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Ε, ευχαριστώ που είστε παρούσα. Ε, πρώτα θα ακούσουμε μια δεκάλεπτη παρουσίαση από την επιλεκτήσα υποψηφία κυρία Ντεμπόλ και μετά θα ακολουθήσει μια πρώτη σειρά ερωτήσεων από τους συντονιστές και από οτιδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και μετά, αν μας επιτρέπει ο χρόνος και αν είναι αναγκαίο, μια δεύτερη σειρά ερωτήσεων. Σας εύχομαι, ένα, σας εύχομαι θερμός καλώς ορίσατε, κυρία Τζεμπόλ. Εάν είστε έτοιμες και έτοιμοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να παρακολουθήσετε τα όσα θα αναπτύξει η κυρία Τζεμπόλ, θα της δώσω 10 λεπτά και μετά θα μπορέσετε να θέσετε ερωτήσεις. Καλώς ήρθατε πρώτη φορά εδώ στην Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την παρουσίασή σας αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρίες και κύριοι σαν υποψηφία για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της Europol σας ευχαριστώ που μου δώσατε την δυνατότητα να παρουσιάσω τον εαυτό μου και να εκφέρω τις απόψεις μου για θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας και για τη Europol στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Θα μπορούσα να έχω παρακαλώ την πρώτη διαφάνεια, λέει η κυρία Ντεμπέλ. Libe takes full responsibility for this. <laughs> <laughs> Given it's your <laughs> there we go. Here we are. Yes. I will give you my reflections on a safer Europe and the role of Europol. Θα σας μεταφέρω τις απόψεις μου για την ασφάλεια της Ευρώπης. Η επόμενη λοιπόν διαφάνεια. Αυτά σας δίνουν μία εικόνα των αρμοδιοτήτων τις οποίες πρέπει να έχει μία αστυνομική και κατασταλτική αρχή. Είμαι δικηγόρος, είμαι νομικός μάλλον. Ξεκίνησα σε μια τοπική αστυνομία και μετά έγινα ε, επιθεωρήτρια στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία Η βασική αρχή που με έχει οδηγήσει μέχρι τώρα είναι ο σεβασμός για την ανθρώπινη ζωή, ο σεβασμός για τη δημοκρατία και τους κανόνες του δικαίου. όπως επίσης σεβασμός και διαφάνεια απέναντι στην πολιτική εξουσία, απέναντι στο προσωπικό των αστυνομικών αρχών και τους πολίτες. Θα πρέπει να σεβαστούμε τους ρόλους των διαφορετικών διακριτών εξουσιών επίσης ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες και τις ε, επενδύσεις για νέους εξοπλισμούς των αστυνομικών αρχών. Εδώ θα σας μεταφέρω τις απόψεις μου για τις απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε επίπεδο ασφαλείας, τις προτεραιότητες της Europol και τον ρόλο τον οποίο πρέπει να αποκτήσει η Europol. Ε, υπάρχουν πολλές περίπλοκες μορφές τρομοκρατίας όπως το έγκλημα παραμένει βασική ανησυχία για τους Ευρωπαίους πολίτες και οι Ευρωπαίοι πολίτες αναγνωρίζουν ότι το κυβέρνο έγκλημα είναι μια σημαντική απειλή. Οι μελέτες δείχνουν επίσης ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να υπάρξει μια αύξηση της κατανομής και ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης ανάμεσα τις διάφορες χώρες σε θέματα τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος. Οι πληροφορίες ανταλλάσσονται όλο και περισσότερο και αυτό είναι θετικό, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό. Η Europol και οι εθνικές κοινότητες ασφαλείας θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις αυτές. Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη θα συνεχιστούν, θα πάρουν διαφορετική μορφή Γι' αυτό η Europol θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για το μέλλον και θα πρέπει να είναι σε θέση να υπερβεί το παρόν πλαίσιο και να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές απειλές από πλευράς τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος. Για να μπορέσει η Europol να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουμε. Είναι μια ισχυρή, σύγχρονη οργάνωση και είναι έμπιστος εταίρος για όλους και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και τον προκάτοχό μου, διότι πραγματικά μετέτρεψε την Europol σε μια σύγχρονη αστυνομική αρχή όπως την βλέπουμε σήμερα. Θέλω να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και να μπορέσει να καλύψει τις ανησυχίες των πελατών της. Ως εκ τούτου η βασική μου προσπάθεια, ο βασικός μου στόχος θα είναι οι κεντρικοί πελάτες αν θέλετε, είναι οι ανησυχίες και οι ανάγκες των κρατών μελών. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των κρατών μελών. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη, προβλέπεται στον κανονισμό μας, και θα πρέπει να γνωρίζουμε και να κατανοούμε καλύτερα το τι επιθυμούν οι πελάτες μας αυτοί, να μπορούμε να αξιολογούμε και να μαθαίνουμε από τις ανάγκες αυτές και φυσικά να είμαστε ικανοί και στην απάντησή μας. Αυτό περιλαμβάνει ότι θα πρέπει να ισορροπήσουμε τις ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προτεραιότητες των, τις εθνικές των κρατών μελών. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η διαχείριση της πληροφόρησης και ενημέρωσης μέσω της καινοτομίας και της πρόβλεψης γιατί είναι αυτό ε, καθοριστικό. Η Europol θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργαστεί όλες τις πληροφορίες τις οποίες παίρνει και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να διαχειριστεί τις νέες πληροφορίες τις οποίες θα λάβει αύριο μέσω drone κτλ. Γι' αυτό λοιπόν η Europol θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες μορφές ενημέρωσης και στις νέες σκέψεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί η απαιτούμενη προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ήδη φτάσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί από πολύ κοντά τις ψηφιακές ε, εξελίξεις και να προβλέπει τις νέες καταστάσεις και στα πλαίσια του καθεστώτος προστασίας δεδομένων και στα πλαίσια του σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων. Τώρα μπορεί να το κάνει μόνη της αυτό η Europol. Όχι βέβαια. Η Europol θα πρέπει να λειτουργήσει από κοινού με τους εταίρους της, άλλες υπηρεσίες, να υπάρχει δηλαδή μια συνεργατική στάση απέναντι στις υπόλοιπες κοινοτικές υπηρεσίες. Για να μπορέσει να εφαρμόσει τις προτεραιότητες αυτές η Europol θα πρέπει να είναι ανθεκτική θα πρέπει να είναι ευκίνητη για να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις ανάγκες της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό. Η Europol θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και τους νέους κινδύνους, να στηρίζει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών και να λειτουργήσει προληπτικά, να είναι στραμμένη στο μέλλον θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι μελλοντικέ απειλές, θα πρέπει να δούμε τι συνέπειες των μελλοντικών αυτών απειλών, θα πρέπει να δούμε πώς οι δυνάμεις ασφαλείας θα πρέπει να προετοιμάζονται για το μέλλον και πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι και ε, κέντρα πρόβλεψης των επερχομένων αλλαγών. Να δούμε ποιο είναι το πολιτικό πλαίσιο και ποιο είναι το πλαίσιο ασφαλείας μέσα στο οποίο κινούμεθα. Έτσι θα μπορέσουμε να δει οι αστυνομικές δυνάμεις στη συγκεκριμένη περίπτωση περισσότερο αντέδρασαν παρά προέβλεψαν και κανένας δεν προείδε τις δυνατότητες που είχαν ε, ε, οι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος να εκμεταλλευτούν τα, τα παιδιά. Έπρεπε να το είχαμε προβλέψει αυτό πρέπει να ε, απαραίτητο να γίνονται σεβαστά. Έχουμε το σύστημα Σιένα, ένα από τα ασφαλέστερα συστήματα μετάδοσης πληροφοριών. Έχουμε τα μέσα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, έχουμε κινητές υπηρεσίες και απαιτείται να έχουμε επίσης και την στρατηγική ικανότητα πρόβλεψης έτσι ώστε να ε, ξελίξουμε τις βέλτιστες πρακτακοσίων μελών, χάρη και στη δική σας προσπάθεια, μπορέσαμε να αναπτυχθούμε. Ε, χάρη σε αυτό η Europol, δεδεμένη οργάνωση η Europol, η οποία θα πρέπει να αναπτύξει την δικτύωσή της ακόμα περισσότερο για να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να είναι ένας αποτελεσματικός και ε, καλός εταίρος στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας πρέπει να ενισχυθεί για να καταστεί πλήρης ε, εταίρος της Επιτροπής ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Θα είμαι στην διάθεσή σας σε όλες τις φάσεις στο μέλλον και θα μπορέσω, ε, εφόσον μου εμπιστεύεστε, να διαχειριστώ σωστά. Ευχαριστώ πολύ. συνάδελφοι. Στον κατάλογο μου έχω κάποιου συναδέλφου στη θέση των βεβαίω, αλλά και συνεισηγητή επί του θέματο. Παρακαλώ. Η... Με ικανοποίησε η συγκεκριμένη παρουσίασή τη, απλή αλλά και έμπλεη περιεχομένου. Έχετε ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα, την οποία εκτιμούμε δεόντως και γι' αυτό δημιουργήσαμε την κοινή ομάδα ελέγχου κοινοβουλευτικού που αποτελείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών μέσω δύο συγκεκριμένων κανονισμών. Θα ήθελα λοιπόν συγκεκριμένα να είπατε ορισμένα στοιχεία μέχρι τώρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτείται να αντιμετωπίσουμε και μία το 17 τον Σεπτέμβριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κυβερνοασφάλεια. Θα ήθελα να μου πείτε τι μέτρα προβλέπετε να λάβετε για να βελτιώσει το 17 τον Σεπτέμβριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κυβερνοασφάλεια. Θα ήθελα να μου πείτε τι μέτρα προβλέπετε να λάβετε για να βελτιώσετε την αποδοτικότητα και την μάχη ε, εναντίον του κυβερνοεγκλήματος. Τι ακριβώς αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω δεδομένου του βιογραφικού σας και επειδή εργαστήκατε στη χωροφυλακή του Βελγίου. Είσαστε Βελγίδα αστυνομικό. Θέλω να ρωτήσω από την βελγική σας εμπειρία, ποια είναι τα σημαντικότερα μαθήματα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τι θα προσφέρετε. Όμως να σας ρωτήσω, τι θα λέγατε, εάν βλέπατε σε κάποια κάτι μέλη και ιδίω κάποιου τομής. γιατί αυτή την παρέα ερώτηση. Σε ένα από τα κράτη-μέλη μας, έγινε μια δολοφονία που προκάλεσε τον αποτροπιασμό όλων μας. Η δολοφονία της δημοσιογράφου Καρβάνα Γκαλήθια. Και η Ευρωπόλ ε, έκανε κρίσει για την έρευνα του εγκλήματος, αλλά τα μέλη της οικογένειας λέγανε ότι η Ευρωπόλ και όλοι εγκαταλείψαν την έρευνα επειδή οι ύποπτε οργανωμένου εγκλήματο, αλλά δεν μπορούσαν να εντυπωστούν οι ευθυντικοί αυτούργοι. Έχετε κάτι να μα πείτε γι' αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Στίβεν από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Ντεμπόλ που είστε εδώ και που μας παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας για το, δράμα, ε, για το μέλλον. Έχω κοινωνικά δίκτυα για να καταπολεμήσει την ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Τι μπορούμε να κάνουμε για να έχει περισσότερο, περισσότερη ε, επίδραση η δράση μας στον ιδιωτικό τομέα και επίσης για τις ιδιωτικές δυνάμεις στην Ευρωπόλ για να συνδράμε τα κράτη-μέλη στις προσπάθειες αποκρυπτογράφησης, αποκωδικοποίησης. Μπορεί δηλαδή να πηγαίνουν εκεί τα κράτη-μέλη και να ζητούν αποκρυπτογράφηση για WhatsApp και Messenger και, τέτοιες, και τέτοια chat με κρυπτογραφημένα μηνύματα. Τι άποψη έχετε εσείς για Στην Επιτροπή για το Οργανωμένο Έγκλημα και την Τρομοκρατία. Ευχαριστώ και για την Γκουε, μάλλον για τους πράσινους, ο κύριος Τερικάμπρας. Sorry. Η κυρία Βίκστρομ από την Άλντε. Παρακαλώ να με συγχωρείτε. Να με... Ε, ελπίζω ότι εδώ έτσι όπως έχω κάτσει περιστοιχισμένη από Βέλγους συναδέλφους δεν υπάρχει περίπτωση να με δείτε, μα είναι τόσο πολύ Βέλγοι σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πολύ διεξοδική παρουσίαση και ήταν επιτέλους ε, μια ευχάριστη αλλαγή να έχουμε τέτοια καλή ενημέρωση για το δύσκολο μέλλον που ξέρουμε ότι περιμένει την Ευρωπόλ. Ξέρουμε όλοι ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία είναι καθοριστική σημασία για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Ξέρουμε ότι η Ευρωπόλ σήμερα είναι εξοπλισμένη, έχει αναλάβει μάλλον ένα, ε, μια ευρύτερη εντολή ε, για τι αρμοδιότητέ τη ε, και να μην ξεχάσουμε ότι και στο μέλλον το κέντρο για το κυβερνοέγκλημα και την καταπολέμηση τη τρομοκρατία είναι υπηρεσίε που ίσω θα δημιουργηθούν σύντομα. Τι προβλέπετε εσύ μετά ως εξέλιξη, μα είπατε ότι δεσμεύεστε για την ενίσχυση τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Το εκτιμώ ιδιαίτερω. Και δεν είναι μυστικό ότι η ομάδα μου, η πολιτική μου ομάδα, η φιλελεύθερη, είμαστε υπέρ αυτού του είδου τη ανταλλαγή πληροφοριών. Και έχουμε τονίσει ότι οι πληροφορίε αυτές σε πολλέ περιπτώσει θα πρέπει να είναι υποχρεωτικέ προκειμένου να ορίσουμε ένα σύνολο πληροφοριών που όλοι μπορούν να το ε, γνωρίζουν εκτός από το να έχουμε 20 διαφορετικά σύνολα. Επίσης, πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των πληροφοριών των 100 μελών, διότι όταν, όταν σκεφτούμε την πρόληψη και την ε, έρευνα ή την ε, πάταξη όλων αυτών των ιδεχθών εγκλημάτων, το σημαντικότερο είναι να έχουμε και ποιοτική πληροφορία αυτό λείπει πολλές φορές. Ήδη νομίζω ότι απαιτείται να πείτε πολλά για να απαντήσετε μόνο και μόνο σε αυτά. Θα σταματήσω εδώ και θα τα πούμε και τις προσεχείς ημέρες. Ευχαριστούμε, Σεσίλια. Έχουμε τρεις ε, έμπειρους Βέλγους συναδέλφους. Όποτε θέλουν λοιπόν να μας ζητήσουν το λόγο. Πέντε! Πέντε είναι, πόπο δυσανάλογη εκπροσώπηση. Είδατε, ήδη έχετε φαν club. Ο κύριος Τερικάμπρας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θέλω να ταράξω τον κατάλογο αγορητών. Οι ε, κυρίες προηγούνταν. Κυρία Ντεμπόλ, συγχαρητήρια. Η ομάδα μου που είναι πράσινη ήφα είναι πολύ ικανοποιημένη για την ε, εκλογή σας. Προς στιγμή έχω μία μόνο ερώτηση. Αναφέρατε σεβασμό για τη διαφάνεια ως ε, στόχο του έργου σας. Νομίζω ότι είναι κοινό μυστικό ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες με την Ευρωπόλ ή τουλάχιστον όχι αρκετέ. Και ότι θα βοηθούσε εάν αρχίζαμε να κατονομάζουμε και να επωνυδίζουμε. Άρα, πώς σκοπεύει να ε, ενισχύσει την διαφάνεια η Ευρωπόλ. Θα αρχίσει η Ευρωπόλ να ε, δείχνει ε, ένα προς ένα τα κράτη-μέλη που δεν συνεργάζονται και να τα θα τα υποχρεώνει να συνεργάζονται. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα οι υπόλοιποι συνάδελφοι που ζήτησαν το λόγο, αυστηρός ε, με τη σειρά που τον ζήτησαν. Ο κύριος Μισελ. βολονταριστική διάθεση. Θα ήθελα να μου πείτε σύμφωνα με την άποψή σας τον χώρο που θα χαρακτήριζα ιδεολογικό. Εγώ δεν σύμφωνο απολύτως με αυτά που είπε η κυρία Γκόμες σχετικά με τον ρόλο σας, αλλά ε, ο οποίος είστε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς, ε, κάποιοι από εμά έχουμε πάρει μέρος ε, που κατά τα άλλα εκθέσατε με πάρα πολύ σαφή τρόπο. Ο κύριος Κοέλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχηθώ την στενότερη δυνατή συνεργασία ανάμεσα στον Διευθυντή, τον εκτελεστικό της Europol και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ρόλος της υπηρεσίας για την υπηρεσία. Δεύτερον, θα πρέπει να διασφαλίσουμε το σωστό επίπεδο ανταλλαγής ενημέρωσης και πληροφοριών. Αντί για περισσότερες ενημερώσεις, θέλουμε καλύτερες μορφές ενημέρωσης. Εμείς ενισχύουμε στην παρούσα φάση το σύστημα Schengen, το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών του συστήματος Schengen και του δίδουμε πρόσβαση και στη Europol. Θέλουμε η Europol να ενημερώνεται τακτικά για οποιαδήποτε στο κέντρο ανάλυσης κινδύνου και πώς πιστεύετε ότι θα διασφαλίσετε τη συνεργασία σας με τις υπόλοιπες αστυνομικές δυνάμεις ε, και ταυτόχρονα πώς βλέπετε τον ρόλο της Europol στα πλαίσια της πρόσβασης στα συστήματα ενημέρωσης. Ο κύριος Λόπες Αγουιλάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποια κενά. Πώς θεωρείτε πώς μπορεί να διασφαλιστεί μια καλύτερη και πιο πλήρη ροή πληροφοριών. Ε, είμαι επίσης βέβαιος ότι θα... Υπάρχουν τέλος πάντων υποψίες ότι η Κίνα ασκεί κατασκοπία, κυβερνοκατασκοπία σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει τρόπος να ε, έρθουν κάποιοι αξιωματούχοι σύνδεσμοι και θα σας εξοικονομήσω λίγο εθνικισμό. Ασφαλώς όμως είμαι υπερήφανος που έχουμε μπροστά μας μια Βελγίδα υποψήφια τέτοιας ποιότητος. Είναι υποδειγματική η σταδιοδρομία της, αλλά βεβαίως είναι και εξαιρετικά τα όσα μόλις μας είπε η ε, φιλοσοφία που διακατέχει τη σκέψη της και που μου φαίνεται επίσης υποδειγματική και σε ό,τι αφορά θέματα ασφαλείας, αλλά και βεβαίως η ε, αυστηρή επαγγελματική της συνείδηση. Αγαπητή κυρία, έχω δύο ερωτήσεις. Θέματα που συζητούνται πολύ στην κοινή γνώμη. Ένας αριθμός ανθρώπων αλλά και πολιτικών σχηματισμών ανακατεύουν μετανάστευση με τρομοκρατία. Η ερώτησή μου προς εσάς που θα είστε υπεύθυνοι της Ευρωπόλ. Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα στα δύο αυτά θέματα, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα, εάν υπάρχει ανάγκη. Ε, δεύτερον, διεξάγεται πολλή συζήτηση, λίγο πολύ παντού, για τα παιδιά των τζιχαντιστών που θα επιστρέψουν από Συρία και Ιράκ. Κάθε χώρα λαμβάνει τα μέτρα της ανεξάρτητα. Θεωρείτε ότι σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπόλ μπορεί να προσφέρει κάποια χρήσιμη υποστήριξη στις δράσεις των χωρών μελών. Ε, ολοκληρώσατε τις ε, παρεμβάσεις των μελών μας. Αντιληφθήκατε και εσείς, ε, κυρία Ντεμπόλ, πόσο είναι το ενδιαφέρον το θέση. Διότι έχουμε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αστυνομική